το οποίο είναι κοινή συζήτηση για την σύνοδο κορυφή των G20 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχουμε δηλώσει του Συμβουλίου και της Επιτροπής ε, για την συνάντηση της 11ης και 12 ης Νοεμβρίου και για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 28 και 29 Οκτωβρίου. Επιπλέον, έχουμε την έκθεση Μπερές για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση και τις συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες. Πρόκειται για την ενδιάμεση έκθεση. Και βεβαίως έχουμε την έκθεση ΦΕΙΟ για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλησίου σταθερότητας Ένωσης, ειδικότερα στην Ευρωζώνη. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον κύριο Υφυπουργό των Ολυγία σας ένα λόγο ε, εξ του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, ε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την ευκαιρία που μας δίνει να συζητήσουμε τις προπαρασκευαστικές εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου εν ώψη του επόμενου Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα έχει πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Κεντρικό ζήτημα θα είναι αναμφίβολα η οικονομική διακυβέρνηση. Όπω γνωρίζετε, η Task Force τη οποίας προεδρεύει ο πρόεδρος Φαν Ρομποϊ συνεδρίασε αυτή τη Δευτέρα και ενέκρινε την τελική τη έκθεση που περιλαμβάνει συστάσεις συγκεκριμένα σημαντικές προτάσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε σε ένα ποιοτικό άλμα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα αυτές οι συστάσεις ε, θέλουν να, ε, ε, να τονίσουν την λιτότητα, την πειθαρχία, την διεύρυνση των δυνατοτήτων δράσης σε περίπτωση κρίσης και να ενισχύσουν τους, τους θεσμούς. Όλα αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή σύντομα μέσω της νομοθετικής οδού. Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορέσει να τα εγκρίνει όλα αυτά ώστε να επιτρέψει στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο να προχωρήσουν ε, ταχύτατα σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Κάτι τέτοιο θα ήθελα ένα θετικό μήνυμα όσον αφορά την πρόθεσή μας να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να ανταποκριθούμε στα οικονομικά σε σημαντικές οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι έθεσαν ε, το θέμα άλλων επιλογών που είναι πιο ε, μακριά από αυτές τις τάσεις και ξεπερνούν το πλαίσιο της συνθήκης, όπως ε, η αναστολή του δικαιώματος ψήφου ή η ε, εισαγωγή νέων κανόνων ψηφοφορίας, όπως η αντίστροφη πλειοψηφία. Δεν είναι εύκολα θέματα, ούτε από τεχνικής άποψης, ούτε από πολιτικής και θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας. Ένα άλλο σπουδαίο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αφορά την προετοιμασία της ε, διάσκεψης στο G20 που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει τη θέση της Ένωσης επί τη βάση της προπαρασκευαστικής εργασίας που έγινε εχθές από το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Εν γέννη, ε, είναι σημαντικό η Σεούλ να σηματοδοτήσει μια επιτάχυνση των προσπαθειών που αφορούν την θέση εφαρμογή του πλαισίου για την προώθηση μιας πιο στεναρής, βιώσιμης και έντονης ε, ανάπτυξης. Να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι στην ανάπτυξη. Από το 2008 με την άφηξη της κρίσης και την απάντηση που δόθηκε σε αυτή, δηλαδή μετά από την αύξηση ε, ε, του κύρους της ισχύω στο G20, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η ίδια η φύση πολλών από τις αποφάσεις που είχαν άμεσες επιπτώσεις στους πολίτες μας ε, πέρασε σε διάστημα κάποιων μηνών από το τοπικό εθνικό επίπεδο στο επίπεδο το διεθνές. Παγκοσμιοποίηση μας, μας υποχρεώνει ε, ε, εφ' εξής, να ενεργούμε ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Γνωρίζουμε όλοι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να φτάσει σε συμφωνία για μια νέα συνθήκη που επίσης είχε σκοπό να ενισχύσει το ρόλο της Ένωσης στο διεθνές προσκήνιο. Αυτό μας πήρε 10 χρόνια για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη συνθήκη, αλλά άρχισαν οι τελευταίοι 10 μήνες για να στατοποιήσουμε την ε, σημασία της συνθήκης αυτής. Ε, οι G20 έδειξαν κάποια είχαν κάποιες επιτυχίες από τότε που ξεκίνησα, αλλά νομίζω πως η πιο σημαντική και δύσκολη δοκιμασία είναι αυτή που το περιμένει τους επόμενες εβδομάδες και μήνες, όταν θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό κίνδυνο να χάσουμε το momentum, όπως λέγεται στα αγγλικά, ε, προετοιμαζόμαστε για δύο σημαντικές συναντήσεις και οι δύο στην Κορέα. Η πρώτη σε δύο μέρες είναι η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών και των, ε, γενικών, και των Διευθυντών των Κεντρικών Τραπεζών και η δεύτερη στα μέσα του Νοεμβρίου. Ε, η συμβολή της Ένωσης για μια σταθερή, έντονη και βιώσιμη ε, ανάπτυξη διαφοροποιείται από τη στρατηγική 2020 για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν κυρίως τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πρόγραμμα μεταρρύθμισης του τομέα και της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης. Για το τελευταίο σημείο, στη διάσκεψη κορυφή του Νοεμβρίου, θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα τη Task Force που θα έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Να προσθέσω πω η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη στη διαδικασία peer review στο πλαίσιο του G20. Ως Ευρωπαίοι έχουμε τη συνήθεια και γνωρίζουμε πόσο πολύ μια τέτοιο, ένα τέτοιο είδους εγχείρημα μπορεί να αποδειχθεί ενδιαφέρον και χρήσιμο. Ο καθής πρέπει να παίξει το ρόλο του βέβαια, να αποδείξει καλή βούληση, να συμβάλλει στο πλαίσιο για την ανάπτυξη, framework for growth. Η μάχη δεν δίνεται μόνο σε μια φορά, αλλά πρέπει διαρκώς να είμαστε σε επαγρύπνηση, μέρα με την ημέρα. Ε, κατά τα λοιπά, ενώ η εργασία των τεχνικών ε, οργάνων όπως το Financial Stability Board, το οποίο ε, γίνεται ο Μάριο Ντρόγκη, προχωρά θετικά και ιδιαίτερα η προσανατολισμός του ακολουθεί την σωστή κατεύθυνση για να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να τηρήσουν τις υποχρεώσεις, τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν πέρυσι στο Πίτσμπουργκ ώστε το νέο νομισματικό ταμείο να είναι πιο αντιπροσωπευτικό και να αντανακλά την νέα διεθνή ε, κατάσταση με μεγαλύτερο ρόλο για τις αναδυόμενες οικονομίες. Αλλά θα είμαι σαφής εδώ, δεν μπορούμε να περιμένουμε η Ευρώπη μόνη της να κάνει όλες τις υποχωρήσεις στο θέμα. Όλες οι προηγμένες χώρες θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν. Ήδη εμείς δείξαμε διαθεσιμότητα συγκεκριμένα όσον αφορά την αντιπροσώπευση, τη διακυβέρνηση αλλά και των ε, ποσοστών και νομίζω πως αποτελεί αυτό μια καλή βάση για να φτάσουμε σε συμβαστική λύση. Να μην πει κανείς λοιπόν πως η Ευρώπη αν δεν κινηθεί τίποτα στο θέμα αυτό. Τώρα, ως Ένωση έχουμε ε, μεταξύ μας διαπραγματεύσεις για όλα αυτά και για διάφορες, ε, διάφορα θέματα κλειδιά για τους όρους αναφοράς για την επαφή, τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών του G20 που θα γίνει αυτή τη βδομάδα. Και αυτό έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι όχι μόνο να μιλούν με μια φωνή, αλλά επίσης να εστιάσουν στην υπεράσπιση και την προώθηση όσων είναι τα πιο σημαντικά του συμφέροντα. Η Προεδρία και η Κομισιόν θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να υπερασπιστούν αυτά τα συμφέροντα που προκύπτουν από την κοινή μας θέση η οποία με τη σειρά της είναι αποτέλεσμα εργασίας πολλών μηνών και όλων των κρατών μελών. Τώρα, για το κλίμα. Πρόθεσή μας ε, δεν είναι να έχουμε μια εισβάθος συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί το Συμβούλιο για το Περιβάλλον στις 14 Οκτωβρίου που μας πέρασε υιοθέτησε ένα συγκεκριμένο κείμενο συμπερασμάτων που ορίζει την ευρωπαϊκή θέση. Ε, καθίσατε όλο ένα και πιο επίγον να δημιουργήσουμε, να θεσπίσουμε ένα καθεστώς πολύ φιλόδοξο για το κλίμα μέχρι το 2012 και με το στόχο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει μια σταδιακή προσέγγιση με βάση το Κιώτο και τη διάσκεψη της Κοπεχάγης. Ένα διεθνές πλαίσιο πλήρες, δεσμευτικό που θα λαμβάνει υπόψη τους πολιτικούς προσανατολισμούς που ε, καθορίζονται στο τελικό κείμενο της Κοπενχάγης. Η διάσκεψη του Κανκούν θα πρέπει να φτάσει σε ένα ισόρροπο αποτέλεσμα που θα λαμβάνει υπόψη τα ανησυχίες όλων των μερών και θα θεσμοθετεί τις προόδους που έχουν ήδη σημειωθεί μέχρι σήμερα. Εμείς εκφράσαμε την προτίμησή μας για ένα μέσο ενιαίο δεσμευτικό και νομικό που θα περιλαμβάνει και θα βασίζεται μάλλον στο πρωτόκολλο του Κιώτου. Βεβαίως προβλέπουμε μια δεύτερη περίοδο ε, δέσμευσης με βάση το πρωτόκολλο του Κιώτου αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ε, τη βάση μιας μεγαλύτερης δέσμευσης που θα προσυπογράψουν όλες οι μεγάλες οικονομίες και όπου θα μεταφράζεται η αποτελεσματικότητα της διεθνούς δράσης και θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εγγυηθούμε επιγόντως την ακαιρεότητα του περιβάλλοντος. Θα ήθελα τώρα σύντομα να σας αναφέρω την προετοιμασία για την ευρωπαϊκή θέση εν ώψη της διάσκεψης κορυφής με τη ΣΥΠΑ, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Ήταν η πρώτη φορά που η προετοιμασία διάσκεψης κορυφής με τους εταίρους κλειδιά ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται σε επίπεδο αρχηγών κατών και κυβερνήσεων με βάση τα όσα αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Ε, η ιδέα είναι να βελτιώσουμε τις σχέσεις με τους εταίρους μας χωρίς να θέλουμε να, να προκαταβάλουμε τα πορίσματα. Θα σας πω ε, πώς προετοιμάζεται αυτή η επερχόμενη διάσκεψη ε, κορυφής. Διάσκεψη κορυφής με τις ΕΠΑ βάσει κάποιων θεμάτων κλειδιών. Ενίσχυση Τη ε, διατλαντική συνεργασία, που είναι βασικός φορέας για την επεξεργασία ε, αποτελεσματικών λύσεων στις κοινέ προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Την επαύριο δε της ε, διάσκεψης του G20, η διάσκεψη κορυφή Ευρώπη ήπα θα είναι ένα σημαντικό φόρουμ ώστε να μιλήσουμε και να καταγράψουμε τα όσα έγιναν όσον αφορά τα οικονομικά θέματα αλλά και να αναζητήσουμε κοινή προσέγγιση απέναντι σε αναδυόμενες οικονομίες η διάσκεψη κορυφή αυτή θα επιτρέψει να ξεκινήσει και πάλι το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο που θα αποκτήσει ίσως κάποιες περισσότερες αρμοδιότητες παρά να είναι ένα απλό μέσο ρυθμιστικό. Ε, μέτρα μπορούν να ληφθούν επί τη βάση μιας ενισχυμένης εντολής για διάφορα θέματα οικονομικά ή και απασχόλησης. Θα προετοιμάσουμε επίσης τη διάσκεψη της Κανκούν ένα σημαντικό μήνυμα από πλευρά των, των Αμερικανών εταίρων έχει φτάσει. Άλλα θέματα διεθνούς πολιτικής, ε, όπως το Σουδάν και το Ιράν, θα είναι επίσης στην ε, ημερήσια διάταξη. Για την Ουκρανία προβλέπεται απόψε συζήτηση με την ΥΠΑ το πρόσωπο και θα μου επιτρέψετε να μην πω περισσότερα από αυτού. Για τη Ρωσία και θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη στήριξή μα για την εταιρική σχέση για τον εξυγχρονισμό που θα επιτρέψει να ενισχυθεί η συνεργασία μα σε όλου του τομεί και κυρίω στου τομεί κλειδιά όπω η καινοτομία και η ενέργεια. Αυτά, Πρόεδρε, κύριε, ε, Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, τα θέματα τα, λοιπόν στο Συμβούλιο, όπως σας είπα, για την επόμενη εβδομάδα είναι πολλά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας κάνατε. Πολύ σημαντική για μας. Καλωσορίζω τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο κύριε Μπαρόζο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, Πρόεδρε του Συμβουλίου, αξιότιμα μέλη. Συζητούμε καταρχήν τα θέματα τα οποία θα συζητήσει την επόμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα συγκεντρωθώ, θα εστιαστώ στα πιο σημαντικά κατά την άποψή μου θέματα. Οικονομική διακυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά τι εξωτερικέ μα δράσει τη συνοκορφή με τι ΗΠΑ και με τη Ρωσία ασφαλώ, που είναι κρίσιμε, ε, θα αναφερθώ και στην συνοκορφή στη Σεούλ του G20 και την διάσκεψη κλιματική αλλαγή του Κανκούρ. Η αναμόρφωση της ε, οικονομικής διακυβέρνησή μα είναι απολύτως απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε αξιοπιστία και οικονομική ανάκαμψη. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν έχει πάρει πολύ στα σοβαρά αυτό το θέμα. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Κομισιόν τον περασμένο, ε, μήνα ε, χαρακτηρίζονται από το επίγον της αντιμετώπισης της κρίσης μέσα, μέσα στην πραγματικότητα τη σημερινή. Θέλουμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύ στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής μέσω συντονισμένης ε, ε, μακροοικονομικής εποπτείας και ε, αντιμετώπισης των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Το λέμε δηλαδή συχνά, δημιουργούμε μια πραγματική οικονομική ένωση στην Ευρώπη. Καλωσορίζω την πρόθεση, την προσοχή του Κοινοβουλίου σε αυτές τις προτάσεις. μια γρήγορη συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση θα μας επέτρεπε να προχωρήσουμε σε πράξη οι κανόνε αυτοί θα έπρεπε να αρχίσουν να εφαρμόζονται από τα μέσα του επόμενου έτους. Θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε να πετύχουν αυτού τους ε, στόχους και να δώσουν συνέχεια επιγόντω σε αυτή την ατζέντα. Έχουμε κινηθεί σε πιο ισχυρή ε, ε, ομοφωνία, σε πιο ισχυρή συμφωνία για πολλά από αυτά τα θέματα με βάση τα πορίσματα ε, της ε, Task Force υπό την προεδρία του κ. Φαν Ρομπέι. Όταν τα ολοκληρωθούν αυτές οι συζητήσει και ληφθούν οι αποφάσεις, το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα έπρεπε να είναι το εξής. Ένα όραμα για μια οικονομική διακυβέρνηση που θα είναι πολύ πιο σφαιρική και πιο συντονισμένη με την ανάγκη πρόληψης των προβλημάτων και που θα βασίζεται πολύ περισσότερο στην χρήση κυρώσεων όμως να καταστήσω σαφές το εξή. Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να αντιπροσωπεύει μια πραγματική αλλαγή σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση προς όφελος των πολιτών μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ε, θα πρέπει να βγάλουμε τα διδάγματα που πρέπει από αυτή την κρίση. Ορισμένα θέματα ακόμα εκκρεμούν. Ένα από αυτά είναι πώς θα αντικαταστήσουμε τον σημερινό τρέχοντα μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσης που συμφωνήθηκε το Μάιο με ένα μηχανισμό πιο μόνιμης φύσεως ε, όταν θα λήξει ο τρέχον μηχανισμός το 2013. Θα πρέπει να αποφύγουμε την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων στο μέλλον, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να είμαστε προετοιμασμένοι για κρίσιμε εξελίξει όπως αυτές των τελευταίων μηνών. Θα πρέπει να έχουμε ένα μόνιμο μηχανισμό που θα προλαμβάνει τέτοιου είδους κρίσει στο μέλλον. Η Κομισιόν έχει λάβει γνώση των απόψεων των κρατών μελών που ε, επιθυμούν μια αλλαγή στη συνθήκη. Για τέτοιου είδους αλλαγές χρειάζεται βέβαια ομοφωνία όλων των κρατών μελών. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν εστιάζεται στην ουσία τι εννοώ. Σχεδιάζουμε ένα μόνιμο μηχανισμό που θα παρέχει αναχώματα σε κρίσιμες στιγμές, μειώνοντας τον ηθικό κίνδυνο και εξασφαλίζοντας ότι αυτός ο μηχανισμός θα χρησιμοποιείται ως ε, τελευταία λύση. Όταν υλοποιηθεί πλήρως, το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας θα είναι αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι ένα σύστημα που θα έχει κίνητρα στα κράτη, θα δίνει κίνητρα στα κράτη-μέλη να ακολουθούν υγιείς ε, δημοσιονομικές ε, πολιτικές και ε, θα ελέγχονται ε, από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Με λίγα λόγια, βγάζουμε διδάγματα και γι' αυτό το λόγο ετοιμάζουμε ένα σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης τελείως καινούριο σε σχέση με την κατάσταση πριν από την κρίση. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε αυτό το σύστημα σε πολύ πιο υγιή θεμέλια. Το παρελθόν μας στο, στην οικονομική διακυβέρνηση θα μας ε, δώσει την ευκαιρία να πάμε στην G20 που είναι πολύ επίκαιρη και κέρια συνάντηση έτσι ώστε να συντονίσουμε οικονομικά την δράση μας σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο έτσι ώστε να πετύχει αυτή η συνάντηση του G20. Τι θέλουμε να πετύχουμε. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα του G20 έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης μέσω συλλογική δράσης. Τώρα περνάμε σε μια καινούργια φάση και σε αυτή τη φάση θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως οι παγκόσμιες ανισορροπίες ανησυχούν όλου μας και όλες οι μεγάλες οικονομίες έχουν ε, τμήμα της λύσης. Δεν θα πρέπει να αγνοούμε την πραγματικότητα ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι πολύ σημαντικές. Δεύτερον, θα πρέπει να αναλάβουμε δράση και στα διεθνή οικονομικά όργανα. Θα πρέπει να ανασχηματιστεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, και οι άλλοι διεθνείς οργανισμοί και φορείς. Με την υποστήριξή σας ε, αυτή τη στιγμή προβαίνουμε και σε μεταρρύθμιση του δικού μας οικονομικού συστήματος ε, χρηματοοικονομικού συστήματος και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τονίσατε την ανάγκη να πετύχουμε. Πρέπει να διατηρήσουμε την ορμή μας και στη συνάντηση του G20. Έχουμε ήδη πετύχει πρόοδο, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχιστεί και στην υλοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μείνει προσιλωμένη στο στόχο τη. Μεταρρυθμίσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα θα, θα δούμε και άλλους τρόπους έτσι ώστε ο χρηματοοικονομικός τομέα να συνεισφέρει επαρκώς ε, στην σταθερότητα σε, κοινοτικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, η ατζέντα του G20 επίσης περιλαμβάνει και την ανάπτυξη ως σημείο της. Θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας διότι η Κομισιόν ήταν πάντοτε ε, υπέρ τέτοιων δράσεων. Η ατζέντα του G20 θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις αναπτυσσόμενες χώρες και να τις βοηθάει. Ταυτόχρονα θα πρέπει οι αναδυόμενες οικονομίες να μπουν στο πλαίσιο παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με, τις, με τους στόχους της ε, αναπτυξιακής πολιτικής και με συντονισμό. Την προηγούμενη φορά που μίλησα στο Στρασβούργο ε, με τον κύριο Μπάνκι Μουν μου το ανέφερε ρητά και χαίρεται που η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ατζέντα του G20. Τέλος, το G20 θα πρέπει να ε, ηγηθεί στην ε, πρόωθηση της, ατζεν, της εμπορικής ατζέντα. Ε, θα πρέπει η συνάντηση αυτή να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε και να καταλήξουμε στις συνεδριάσεις της Δόχα. Τώρα, σε, ε, ε, στην πορεία προς το Κανκούν έχω να σας πω το εξής. Θα πρέπει να παραμείνουμε εστιασμένοι στους στόχους μας. Να είμαστε ε, φιλόδοξοι για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Ασφαλώς και θα πρέπει να κινηθεί η παγκόσμια διαδικασία και δεν είναι εύκολο. Ορισμένοι μας συνεργάτες και εταίροι αργούν. Έχουν επιβραδύνει αντί να επιταχύνουν. Όμως, μην ξεχνάμε ότι ενδιάμεσα εμεί εφαρμόζουμε ένα πολύ αποτελεσματικό, το πιο αποτελεσματικό σύστημα μείωση των εκπομπών στον κόσμο. Και αυτό είναι το βασικό μα ατού. Όσο πιο φιλόδοξο σύστημα ε, εφαρμόζουμε, τόσο πιο ισχυροί γινόμαστε. Είμαστε πρώτοι σε συνένεση ανάμεσα στην Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Οπότε στο Κανκούν ε, ας ε, εστιαστούμε στην ουσία και όχι στους τύπους. Ας πάμε με αποφασιστικότητα. Το Κανκούν μπορεί να μην είναι το τέλος ε, της, ε, του αγώνα, του δρόμου, αλλά μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική, ένα, σημαντικό στάδιο. Ε, θα πρέπει ο στόχος μας να είναι μέτρα, συγκεκριμένα μέτρα δράσης που θα επαναφέρουν την εμπιστοσύνη στη διαδικασία και θα μας οδηγήσουν πιο κοντά στο στόχο μας. Γι' αυτό το λόγο μίλησα στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα. Είπα ότι θέλουμε μια ρεαλιστική, ισορροπημένη θέση που θα μα ε, σπρώξει προ τα μπροστά χωρί να ε, δημιουργήσει μη ρεαλιστικέ προσδοκίε. Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί της διαδικασίας αυτή, να ε, δείξει πώ το Κανκούν μπορεί να μα προχωρήσει με συγκεκριμένε δεσμεύσει. Και κάνοντα σαφέ ότι η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να είναι παράδειγμα η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναπτυχθεί περισσότερο φέτος από ό,τι είχε προβλεφθεί. Όμως η ανάκαμψη ε, δεν έχει εδρεωθεί ακόμα. Ε, δεν ε, μπορούμε να επαναπαυθούμε, διότι η ανεργία είναι πολύ ψηλή ακόμα. Στους περασμένους μήνες αντιμετωπίσαμε σημαντικές προκλήσεις. Αυτό άλλωστε το αναφέρει και η έκθεση την οποία θα συζητήσετε, η έκθεση Μπερές. Ε, χαίρομαι για την ε, φιλοδοξία και την συνένεση, την ευρία συνένεση για αυτά τα θέματα στο Κοινοβούλιο. Όμως όλοι γνωρίζουμε πως η ανεργία είναι πολύ ψηλή, οι κρατικές ε, δαπάνες μειώνονται, οι πολίτες μας ανησυχούν. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Γνωρίζουμε επίσης ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν έχουμε βρει απαντήσεις. Έχουμε προτείνει ορισμένα σημαντικά νομοθετικά κείμενα, κείμενα για την οικονομική διακυβέρνηση. Έχουμε την Ευρώπη 2020. Είναι μια στρατηγική ανάπτυξη. Το επαναλαμβάνω αυτό. Ανάπτυξη. Εφύση ανάπτυξη. Αυτή είναι η απάντηση. Και αυτό το αναφέρει και ο κ. Φέιο στην εξαιρετική του έκθεση. Έχουμε προτείνει πολλά μέτρα εποπτείας των χρηματοοικονομικών αγορών. Έχουμε κάνει προτάσεις χρηματοοικονομικής εποπτείας. Αν πριν από δύο χρόνια μα ρωτούσαν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για ένα τέτοιο υποπτικό σύστημα, ε, θα απαντούσαμε όχι. Σήμερα όμω είναι δυνατόν. Ε, ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση για όλες τις διαστάσεις. Συμφωνία, για παράδειγμα, που επήλθε χθε στο Συμβούλιο για την πρόταση της ε, για τα hedge funds, ε, τα μια στάθμιση κινδύνου η πρόταση αυτή θα περάσει από το Κοινοβούλιο έτσι ώστε τελικά ε, να υιοθετηθεί αυτός ο κανονισμός τον οποίο περιμέναμε πολύ καιρό. Και πάλι θα είμαστε πρώτοι, θα ηγούμαστε σε όλο τον κόσμο για αυτό το θέμα. Ε, αλλά σημειώνουμε πρόοδο και σε άλλα ζητήματα. Πρέπει να δούμε για την πραγματική οικονομία. Να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για τι εργασίε του περί τη καινούργια οδηγία για την καταπολέμηση καθυστερημένων πληρωμών σε οικονομικέ συναλλαγέ. Αυτή η οδηγία θα δώσει μεγαλύτερη ε, ε, προστασία σε πιστωτές όπου τις περισσότερες φορές είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, θα πρέπει μέσα να γίνονται σε 30 μέρες, αλλιώς θα γίνονται με ε, τόκο. Ξέρετε πόσο το περιμένουν αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο μας. Οι προτάσεις μας θα πρέπει να υιοθετηθούν μέχρι τέλους, αλλά ήδη δίνουν αποτελέσματα καρπούς. Στόχος είναι να βγούμε από την κρίση και μέσω της ανακάμψης να ξαναπετύχουμε ε, τους ρυθμούς ανάπτυξης που θα μειώσουν την ανεργία και ε, που θα προσαρμόσουν το κοινωνικό μας κράτος στον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Παρόζο. Καλημέρα σε όλους. Θα δώσουμε τώρα το λόγο για τέσσερα λεπτά στην κυρία Περβάνς Μπερές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, η οικονομική, η χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο εδώ και αρκετά πλέον χρόνια θα κοστίσει 60 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμια κλίμακα, δηλαδή ένα, μια ποσοστιαία μονάδα ετησίως. Θα μεταφραστεί σε ένα ποσοστό ανεργίας στη δική μας Ευρωπαϊκή Ένωση του 11% μέχρι το τέλος του έτους μεταφράζεται τη στιγμή όπου ο πόλεμος, ε, ο νομισματικός ε, ε, μένεται θα μεταφραστεί σε μια κατάσταση κινδύνου ε, στην ε, νιωστή, όπως λένε οι οικονομολόγοι μας. Εν ώψη αυτής της κατάστασης κάνω έκκληση στο Κομισιόν, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για να πω ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε γύρω από την προστιθέμενη αξία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, του ευρωπαϊκού σχεδίου και έχουμε και να σας θυμίσω πως φέρουμε συλλογική ευθύνη και σε επίπεδο σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουμε να θέσουμε μια στρατηγική σε κίνηση ώστε να μας επιτρέψει να είμαστε ισχυροί στο εσωτερικό της Ένωσης και άρα και στο εξωτερικό. Πρέπει να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις και γι' αυτό χρειαζόμαστε το ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμω, κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή, η οικονομική διακυβέρνηση για μα δεν είναι ένα όραμα είναι ένα μέσο για την εξυπηρέτηση αυτής τη στρατηγικής και γύρω από αυτή τη στρατηγική ορίζουμε τα απαραίτητα μέτρα. Καταρχήν είναι ε, οικονομικά μέτρα. Είναι η φάση της αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών. Με αυτή την κινητοποίηση γύρω από μια στρατηγική για μια ευρωπαϊκή κοινότητα ενέργειας ε, είναι η ανάγκη να κινητοποιηθεί μια πρόταση την οποία εσείς αρνείστε τη φορολόγηση των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Είναι η στιγμή να δημιουργηθεί ένα μεγάλο ευρωπαϊκό δάνειο για να χρηματοδοτηθούν οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Είναι η ανάγκη να εξισορροπήσουμε και πάλι την οικονομία στην Ευρώπη ώστε να είναι πιο ευνοϊκή στην απασχόληση και λιγότερο ευνοϊκή για το κεφάλαιο καθώς και να σέβεται περισσότερο το περιβάλλον. Ανάγκη να συντονιστούν οι εθνικοί προπολογισμοί με τον ευρωπαϊκό ώστε οι προσπάθειε να συγκλίνουν. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, προτείνουμε τη δημιουργία ενός κυρίου ευρώ που θα επιτρέπει πραγματικά να υπάρχει μια αρμονική οικονομική διακυβέρνηση, ισορροπημένη. Επίσης προτείνουμε να μην εστιάσουμε την προσοχή μόνο στην κατάσταση των χωρών που έχουν έλλειμμα, αλλά να την εξορροπήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τις χώρες που έχουν πλεόνασμα. Προτείνουμε επίσης σε μια ενιαία νομισματική ζώνη να διαχειριστούμε ως κοινό αγαθό το χρέος και να μπορέσουμε να προβλέψουμε αμοιβές αμοιβαίο χειρισμό του, του, του χρέους. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και ε, έχουμε, θα πρέπει να οργανωθούμε γύρω από τις ανάγκες των Ευρωπαίων και όχι με μόνο στόχο την οικονομική σταθερότητα. Θέλουμε μεταρρύθμιση της ε, χρηματοπιστωτικής αγοράς που θα ξαναθέσει θέση επιτάπητο στα θέματα της ηθικής που θα είναι θετικά για τη δημιουργία απασχόληση και τις μακροπρο, μακρόπνες επενδύσεις. Καμιά ευρωπαϊκή πολιτική δεν θα ελκύσει τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα καλύτερά μας στοιχεία για να, δώσουμε, να δημιουργήσουμε τη διάθεση στα κράτη-μέλη. Και αυτό δεν θα γίνει μόνο με μια συζήτηση που θα βασίζεται στις κυρώσεις. Έτσι δεν θα τους δημιουργήσετε καμιά όρεξη να κινητοποιηθούν με τα κράτη-μέλη τους οι Ευρωπαίοι και να ε, συσπηρωθούν γύρω από ένα κοινό όραμα. Θέλουμε μια έντονη κινητοποίηση γύρω από την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για να βγουν οι Ευρωπαίοι από την κρίση και να εξασφαλίσουμε πως μεθαύριο στην Ευρώπη όλοι θα έχουν δουλειά, θα, δεν θα ζουν με φτώχεια και θα μπορέσουν εκ νέου να εμπιστευθούν το ευρωπαϊκό όραμα. Ελπίζω, Πρόεδρε ε, της Επιτροπής, ότι θα μπορέσετε να ε, συμφωνήσετε μαζί μας και θα υιοθετήσετε πολλές από τις προτάσεις που έχουμε εδώ εμείς υιοθετήσει στο σώμα. Σας ευχαριστώ κυρία Μπερές και τώρα θα δώσουμε το λόγο για τέσσερα λεπτά στον κύριο Φέιο. Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε της Επιτροπής, Επιτροπερέν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον ε, πολύ θετικό διάλογο τον οποίο είχαμε με την Κομισιόν και με τους εκπροσώπους Συμβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την έκθεση και την κατέστησαν ε, πραγματικότητα. Τους ε, <clears throat> ε ηγητές καταρχήν με τους οποίους αντάλλαξα απόψεις και κατέληξα σε συνενέσεις. Κάτι που ήταν πολλές φορές δύσκολο. Γιατί στο Κοινοβούλιο υπάρχουν πολλές τάσεις. Από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Από αυτούς που θέλουν περισσότερη κυριαρχία, περισσότερη εξουσία. Μέχρι σε αυτούς που ε, υποστηρίζουν τη δημιουργία συγκεκριμένων οργάνων. Όλες οι απόψεις ε, όμως είχαν τον ίδιο στόχο. Στόχος είναι να βρούμε λύσεις στην τρέχουσα κρίση που απέδειξε ότι η Ευρώπη δεν αποκρίθηκε έγκαιρα. Μερικές φορές θα μπορούσαμε να πούμε δεν αποκρίθηκε καν σωστά. Η κρίση απέδειξε ότι πολλές ε, κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διατηρούν ακόμα μια ε, πολιτική που δεν βασίζεται στην πραγματικότητα. Και γι' αυτόν τον λόγο χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που το Κοινοβούλιο προτείνει με τη δική του φωνή. Ορισμένες είναι βραχυπρόθεσμες και άλλες είναι μακροπρόθεσμες. Ο, οκτώ, κυρίως, οκτώ βασικά συστάσεις ε, προτείνουμε. Ε, πολυμερής ε, εποπτεία της μακροοικονομικής ε, εξέλιξη των κρατών μαλλών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να πετύχουμε τους στόχους της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 με στόχο μια Ευρώπη ανάπτυξης ε, με στόχο την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ε, είναι προτάσεις που γίνονται επίσης για την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά το χρέος ενίσχυση της ε, συνεργασίας μέσω της, ε, ε, του Eurogroup στην ομάδα της Ευρωζώνης και ένα μηχανισμό ε, ε, δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Ενίσχυση των μέσων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ε, νομισματικό, οικονομικό και χρηματοοικονομικό ε, τομέα, καθώς επίσης και βελτίωση αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών στατιστικών. Τέλος, καλύτερη εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων. Το Κοινοβούλιο σε όλα αυτά τα θέματα έχει φωνή, ισχυρή φωνή και στόχος μας είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να συντονίσουν καλύτερα θεσμικά τη δράση τους. Μπορούμε να συνεισφέρουμε έτσι ώστε αυτή η λύση να... αυτές οι προτάσεις να είναι καλύτερη λύση σε ό,τι αφορά και την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων ή δυσκολιών. Από εδώ και πέρα η Ευρώπη θα έχει του μηχανισμούς να απαντήσει καλύτερα στο οικονομικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεισέφερε πολύ σε αυτό και θα το κάνει και στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή ξεκινούμε μια νομοθετική συζήτηση για έξι προτάσεις που υπέβαλε η Κομισιόν. Και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη συζήτηση θα υποστηρίξει τη θέση του. Είναι παράξενο που σε ένα πρόσφατο ε, έγγραφο του Συμβουλίου δεν αναφέρεται η θέση του Κοινοβουλίου και ο διάλογος που έλαβε χώρα μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Όμως να πω το εξής, το Κοινοβούλιο έχει θέση, πάει για θέση και τη διατηρεί παρόλες τις διαφορές μας. Είμαστε υπέρ μια ισχυρή Ευρώπης, μια καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση με μεγαλύτερη ανάπτυξη <clears throat> και μικρότερη ενέργεια. Σας ευχαριστώ κύριε Φέγε. Το λόγο έχει τώρα η συνάδελφος Μάρτα Αντρέασεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στην γνωμοδότησή μου για την έκθεση του κυρίου Φέγε για το πλαίσιο σταθερότητα. Ε, τονίζω τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε σοβαροί στι κυρώσει των κρατών μελών που παραβιάζουν το Σύμφωνο σταθερότητα. Πριν από δύο ημέρε ο Γάλλος Πρωθυπουργό και η Γαλλίδα Καγκελάριο συμφώνησαν να αλλάξουν την συνθήκη για να υπάρχουν ε, αυστηρότερες κυρώσεις για τα κρατη που, αυστηρούν, που απειλούν την ε, σταθερότητα του ευρώ. Επίση, θα πρέπει να υπάρχουν μέσα διάσωσης ε, κάποιου κράτου μέλου στον προπολογισμό και θα πρέπει να δουν ποιο είναι ο αντίκτυπος στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητα της Ένωσης ως αποτέλεσμα του μηχανισμού σταθερότητας. Έχουν αλλάξει λοιπόν οι σχετικές παράγραφοι και δεν αποτελούν πλέον μέρος της γνωμοδότησής μου. Θα ήθελα εδώ πέρα να σας πω πώς αποκηρύσω τη γνωμοδότησή μου κάτω από αυτές τις συνθήκες. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος David Κάζα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι ήταν ε, εξαιρετική αντιμετώπιση της ε, εποπτείας. Βλέπουμε εδώ πέρα πως ε, στις νέες εκθέσεις πρωτοβουλίας για το νέο πακέτο εποπτείας βλέπουμε τους συστημικούς κινδύνους. Από την άλλη, όταν μιλάμε για την ιδέα της οικονομικής διακυβέρνησης, όλοι παραδέχονται πως πρέπει ακόμα να γίνει πολύ δουλειά. Το πρόβλημα στο Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη είναι πω μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε άλλε χώρε, οπότε πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ενθαρρύνουμε τη σοβαρή αναγνώριση των κανόνων επί των οποίων έχουμε ήδη συμφωνήσει για να είναι σταθερά τα κράτη-μέλη και οικονομικά και στα δημόσια οικονομικά τους. Προφανώς ε, χρειάζεται επίσης ε, δουλειά για την ε, οικονομική διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Κορέα, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, όλοι αναγνωρίζουμε ότι απέτυχε ο έλεγχο ο μακροοικονομικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα τα δημοσιονομικά πλαίσια και τα σορευόμενα κρατικά χρέη. Ε, θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι προτάσεις Μόντι και Γκρέκ όσον αφορά τις ε, διασυνοριακές πληρώσεις, ε, πληρωμές, συναλλαγές, να διευκολυνθούν οι online συναλλαγές για να μπορέσει να δοθεί εμπιστοσύνη, να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στους καταναλωτές και να βελτιωθεί η οικονομία. Θα πρέπει επίσης να έχουμε ε, υπεύθυνου προπολογισμού, αλλά και ακατάλληλους και αξιόπιστου δείκτε. Ε, οι δείκτε απασχόλησης θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη στο σύστημα υποπτία. Οι δείκτε ε, για τη στρατηγική 2020 δεν μπορούν επίσης να μείνουν πίσω. Θα πρέπει να μας δείχνουν κοινέ ευρωπαϊκέ προοπτικές και να δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογή διαφόρων μέσων για την υπεράσπιση της Ευρώπης απέναντι στην κερδοσκοπία. Ε, η δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου βρίσκει την στήρι... μας βρίσκει σύμφωνος ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τους ε, κερδοσκοπικούς χειρισμούς ε, στην αγορά. Η έκθεση ΦΕΙΟ είναι πολύ ικανοποιητική, μπόρεσε να φτάσει σε ένα πλούσιο κείμενο, πολύ ισόρροπο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κορέιρα Κάμπος και τώρα για μια σύντομη παρέμβαση θα πάρει το λόγο ο κύριος Μάρτιν Σούλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εάν δείτε τον κατάλογο των ομιλητών, βεβαίως φαίνεται ο Ραμόν Γιαουρέγγι ως επόμενος ομιλητής. Πριν όμως λάβει τον λόγο, θα ήθελα να μου επιτρέψετε ως πρόεδρος της ομάδας μας να ανακοινώσω πως ο κύριος Γιαουρέγγι ορίστηκε σήμερα υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας, οπότε είναι τιμή για την ομάδα μας και θα ήθελα να τον συγχαρώ. Ωραία, ευχαριστώ. Και δίνω το, λόγο στον αξιότιμο συνάδελφο Υπουργό Γιαουρέγγι και πολλές ευχές από μέρους όλων μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Μάρτιν. Φίλε μου, ένα λεπτό έχω μόνο στη διάθεσή μου να σας πω ότι πιστεύω πως η Ευρώπη αυτούς τους ε, μήνες έκανε σημαντικά βήματα στην οικονομική διακυβέρνηση. Ε, προχτές ε, η σύνος κορυφής όμως μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας έδωσε μια καινούρια έκανα ε, ε, ένα ακόμα βήμα που είναι η δυνατότητα αλλαγή των ε, συνθήκων κάτι που είναι ένα παράθυρο, μια ευκαιρία για μας οι ευρωπαϊστές ζητούμε η οικονομική διακυβέρνηση που πρέπει να οικοδομηθεί να συνοδευτεί από μεταρρυθμίσεις χρειάζονται μεταρρυθμίσεις συνενετικές και η συμφωνία Γερμανίας, Γαλλίας ανοίγει το δρόμο μέσω της, ε, και της έκθεσης ΦΕΙΟ που θα ε, συζητήσουμε ε, να αλλάξουμε το θεσμικό μας πλαίσιο έτσι ώστε η οικονομική διακυβέρνηση να βοηθήσει στην σύγκληση των οικονομιών, στη δημιουργία μιας οικονομίας ανταγωνιστικής που θα αναδιανύμει τον πλούτο όπως ακριβώς ζητούν οι σοσιαλιστές εδώ καιρό. Σας ευχαριστούμε κύριε Γεωρέγγι. Ε, καλή δουλειά, δεν θα έχετε εύκολη δουλειά. Το λόγο έχει ο κύριος Ζώσεφ Ντόλ. Ευχαριστώ. Ναι, όχι ακόμα. Απαντά ο κύριος Ντόλ. Όχι, δεν είναι μέσα στις φιλοδοξίες μου αγαπητοί φίλοι. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το κοινό σημείο ανάμεσα στη ε, διάσκεψη του Συμβουλίου και του G20 είναι να ε, μπορέσουν να γίνουν απαραίτητε προσαρμογέ και μεταρρυθμίσει ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι να βάλουμε τάξη στη δημόσια οικονομία, στην εθνική και στην κοινοτική και στην εισπεράσπιση του νομίσματό μα στο ευρώ απεγειώνοντας το σε εσωτερικό επίπεδο και υπερασπιζόμενοι την αξία του απέναντι στις άλλες, στα άλλα μεγάλα νομίσματα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ε, κυριαρχηθεί από τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή οικονομία. Εμείς στο ΕΛΚ δεχόμαστε με, ε, θετικά τη δημιουργία της, της προτάσης της Τάσχος Φαν που προβλέπει κυρώσεις για τα κράτη που δεν σέβονται το σύμφωνο σταθερότητας. Όμως η δουλειά αυτή θα πρέπει ακόμα να ευαθυνθεί προς την κατεύθυνση της ε, περισσότερης κοινοτικής μεθόδου και της ε, μικρότερης διακυβερνητικής ε, διαχείρισης και χαιρετίζω την δουλειά της Κομισιόν προς αυτή την κατεύθυνση. Να θυμίσω δε στο Συμβούλιο πως αυτό το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να το ξεχνά, είναι πλέον συνομοθέτης και θα παίξει πλήρως το ρόλο του στις μεταρρυθμίσεις στο μέλλον. Όσο περισσότερο εμπλέκεται το Κοινοβούλιο εκ των προτέρων, τόσο περισσότερο θα έχουμε τις πιθανότητες να καταλήξουμε με ικανοποιητικό τρόπο και ζητώ από τον Πρόεδρο Ρομπάι να το, να το ακούσει αυτό. Η Ευρώπη Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να ασχοληθεί με, για, με τη συζήτηση για τη σχετική αξία των νομισμάτων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει πριν το G20. Η Ευρώπη με τους Αμερικανούς εταίρους θα πρέπει να θέσει τις αναδυόμενες χώρες ενώπιον των ευθυνών τους. Το νομισματικό ε, dumping έχει συνέπειες κοινωνικές τις οποίες δεν μπορούμε να αγνοούμε. Θα πρέπει λοιπόν να συζητηθεί η μεταρρύθμιση του διεθνού ε, συστήματο, αλλά και η σταθερότητα των πρώτων υλών, ιδιαίτερα τα τρόφιμα και η ενέργεια καθώς και η παγκόσμια διακυβέρνηση. Για καθένα από αυτά τα θέματα η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει ένα μήνυμα. Το μήνυμα όμως αυτό θα είναι αξιόπιστο, πιστευτό μόνο αν δημιουργήσουμε τα εσωτερικά όργανα διακυβέρνησης και διαχείρισης που θα είναι αποτελεσματικά σε κοινοτικό επίπεδο για την δημόσια οικονομία μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε την παγκόσμια διακυβέρνηση και δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε σε διεθνέ προσκήνιο παρά αν καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια η οποία συχνά δεν είναι δημοφιλής για την εξυγίανση των οικονομικών μας. Και αν τηρήσουμε αυτές τις προτεραιότητες στον αγώνα κατά της, ε, των κλιματικών αλλαγών, ας πούμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Ντόλ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μάρτιν Σούλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα σας αναφέρω μια πρόταση από την δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Συνόδου των ε, G20 στο Pittsburgh στις 24 ε, Σεπτεμβρίου 2009. Έλεγαν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα περιγράφει την πολιτική και την κοινή πορεία για το πώς θα συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή και ισορροπημένη ανάπτυξη την οποία χρειαζόμαστε να δημιουργηθεί μια ενιαία ανάκαμψη η οποία θα δώσει εκείνες τις καλές θέσεις εργασίας οι οποίες χρειάζονται οι λαοί μας. Ωραία. Υποθέτω πως και φέτος θα γράψουν κάτι τέτοια πράγματα στην επόμενη σύνοδο και σε όλες τις σύνοδους. Γι' αυτό ρωτάω τι έχει συμβεί στο έτος ε, το οποίο πέρασε για να δημιουργηθεί αυτή η αηφόρος και διαρκής ανάπτυξη για να δημιουργηθούν αυτές τις θέσεις εργασίας όπως πολύ σωστά περιγράφεται. Αυτό το οποίο δημιουργήθηκε είναι μια φιλοσοφία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πως οι μονομερείς περικοπές των κρατικών προϋπολογισμών είναι πανάκια για τη σταθεροποίηση της Υπήρου. Αντί να σκεφτούμε πως οι επενδύσεις που θα οδηγήσουν την ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για να δημιουργηθούν περισσότερες δουλειές και έτσι θα ενισχυθούν τα έσοδα του κράτους, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε, για να μπορέσουν να κάνουν βεβαίω το έργο τους και να σταθεροποιήσουν τους προϋπολογισμούς τους. Αυτό το οποίο ζούμε είναι μια μανιχαϊστική αντίληψη στην Ευρώπη. Όλα τα έξοδα είναι κάτι κακό, όλοι, όλες οι περικοπές είναι κάτι καλό. Και βλέπουμε στις χώρες που πλήττονται ισχυρότερα, στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα, έχουμε ύφεση και μηδέν ανάπτυξη. Το αντίθετο δηλαδή από αυτό το οποίο περιγράφεται εδώ πέρα ως στόχη Είναι δραματική η εξέλιξη και γίνεται ακόμη πιο δραματική όταν αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν την κρίση, δηλαδή ο κλάδος, ο χρηματοοικονομικός με την άμετρη κερδοσκοπία, καταλήγει και αυτός να μην συμμετέχει στα έσοδα του κράτους π.χ. με το φόρο χρηματοπιστωτικών ε, υπηρεσιών κάτι το οποίο βεβαίω δεν θα περάσει από τις ε, G20 και βεβαίως δεν θα περάσει γιατί δεν το προσπαθούμε καν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν πέσει σε μια παγίδα η οποία είναι δραματική γιατί μέσω αυτής της αδράνειας των αρχηγών ε, κρατών και κυβερνήσεων ή της δράσης στην λάθος κατεύθυνση θα έχουμε όλο και μεγαλύτερε κοινωνικέ ανισότητες και άνθρωποι που εξεγείρονται στου δρόμου έχουν δίκιο γιατί αυτή η κοινωνική ανισορροπία δεν καταπολεμείται αλλά με τη λάθος αυτή η πολιτική διευρύνεται. Πρέπει να το πει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δείξει στρατηγικές να το καταπολεμήσει. Γι' αυτό προτείνουμε και τον φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και θα δούμε στις εκθέσεις Μπερές και Ποδηματά εάν είμαστε διατεθειμένοι εδώ πέρα Γνωρίζουμε πως είναι δύσκολο, αλλά επιμένουμε να φορολογήσουμε τον τομέα αυτόν, ναι, εάν δεν γίνει σε εθνικό επίπεδο, τότε σε υπερεθνικό. Κυρίε και κύριοι, υπάρχει μια άλλη ανησυχητική εξέλιξη. Αυτό το οποίο έγινε στην Ντοβίλ μεταξύ του κυρίου Σαρκοζή και της κυρίας Μέρκελ. Αντιστρέφει τελείως την θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει καταλάβει ο κύριος Φαν τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί αρχίζει να περιγράφει με την Task Force τι ε, τις μεταρρυθμίσει, απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, αλλά το αποκορύφωμα είναι πως αυτός ο καημένος ο άνθρωπος εργάζεται μυστικά και πριν μπορέσει να υποβάλει οποιαδήποτε ε, ως πρόταση, πάνε στον Ντοβίλ και του λένε ο Νικόλας και η Αγγέλα τα αποφάσισαν όλα στην Τοβίλ. Το γαλλογερμανικό αυτό διευθυντήριο είναι επίθεση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ήμουν εγώ πραγματικά ο Χέρμαν Φανρόπο, θα του το πέταγα στα μούτρα. Δεν είναι δυνατό να το χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα ως, και, να, χρησιμοποιούμε τον Χέρμαν Φανερόμποϊ ως φίλος θα μπορούσαν τουλάχιστον να δουν πως είναι απαραίτητο να, για να αλλάξει η συνθήκη να γίνουν και δημοψηφίσματα και αν κάποιος θεωρεί πω θα δεχόταν κάτι τέτοιο ο κύριο Κάμερον χωρί δημοψήφισμα, κάνει λάθο. Εδώ πέρα λοιπόν θα ανοίξει πραγματικά το κουτί τη Πανδώρα με αυτέ τι εξελίξει. Γι' αυτό το ξαναλέω. Η Ευρώπη πηγαίνει σε λάθο κατεύθυνση και θεσμικά και επί τη ουσία. Ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριο Γκίφερ Χόφστατ. Πρόεδρε, ας ξεκινήσω εκεί που σταμάτησε ο κύριος Σούλτς αν κάποιος ζητήσει αλλαγή της συνθήκης και εμείς θα πρέπει να ζητήσουμε συνέλευση. Ε, διακυβερνητική ενδεχομένως. Ε, δεν έχουμε φτάσει ως εκεί. Ε, θα, αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε επιγόντως ε, είναι η οικονομική διακυβέρνηση, η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, η ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας. Ένα χρόνο μετά την έναρξη της ε, κρίσης του ελληνικού χρέους. Ούτε καν ένας χρόνος δεν έχει περάσει. Το Δεκέμβρη πέρσι ξεκίνησε αυτή η κρίση. Δεκέμβρη του 2009. Λοιπόν, ήρθε ώρα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για αυτό το θέμα. Και έχουμε τρεις προτάσεις αυτή τη στιγμή ε, Α είμαστε σαφείς. Έχουμε την πρόταση της Κομισιόν, την πρόταση της Task Force και από χτέ. και έχουμε από και την πρόταση, την αποκαλούμενη συμφωνία της Ντοβίλ. Και είναι πολύ σημαντικό που το Κοινοβούλιο εξετάζει τις διαφορές ανάμεσα Μάλλον το Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει τις διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις τρει προτάσει και να κάνει τι επιλογέ του. Νομίζω ότι η τη Κομισιόν ε, πριν από μερικές εβδομάδες ήταν ε, καλή, θετική και γενναία. Η Task Force, από την άλλη μεριά, ε, διαφέρει ως προς το, εξή. λέει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει δράση όχι με βάση συστάσεις ε, της Κομισιόν, αλλά με βάση προτάσεις Κομισιόν. Προτάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, συστάσεις μπορούν. Μετά, η Task Force ε, προβλέπει μια πιο μακρόχρονη διαδικασία και αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πρόταση Κομισιόν, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Task Force ε, προβλέπει ένα ημιαυτόματο χαρακτήρα των κυρώσεων και προβλέπει και τον κανόνα αντεστραμμένης πλειοψηφίας ε, που προέβλεπε και η πρόταση Κομισιόν. Τώρα, έχουμε και την τρίτη πρόταση από χτες, πρόταση της Ντοβίλ σίγουρα μια συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας μπορεί να βοηθήσει για τη συζήτηση του θέματος στο Συμβούλιο. Τουλάχιστον αυτό σημαίνει συχνά. Αυτή τη φορά όμως φοβάμαι πως δεν θα γίνει διότι ε, ε, η συμφωνία αυτή στο Συμβούλιο δεν εξασφαλίζει την, το μπλοκάρισμα των ε, προτάσεων περί αυτοματισμού της Κομισιόν. Αντιθέτως, ε, χρειάζεται μια ε, ε, απλειοψηφία για να γίνει κίνηση για την εφαρμογή της, των κυρώσεων. Δηλαδή, καταργείται ο, ο ημιαυτόματος χαρακτήρας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την Ντοβίλ, αλλά εκτός από την παραλία και ορισμένα όμορφα ξενοδοχεία υπάρχει και ένα καζίνο. Τοβίλ. Ε, ίσως δεν θα πρέπει να μιλάμε για την συμφωνία της Ντοβίλ, αλλά για, την, ε, ε, για το συμβιβασμό καζίνο μεταξύ Γάλλων και Γερμανών. Υπάρχει ένα συμβασμό καζίνο, πράγματι. Γιατί τα κράτη-μέλη επιτρέπεται να παίζουν με την ζώνη του ευρώ αν έχουν αρκετή συμφωνία ε, στο Συμβούλιο, όπως ακριβώς έκανε και η Ελλάδα. Faites vos jeux. έτσι είναι. Είναι ένα τυχερό παίγνιο τελικά το, Συμβουλιο, το Σύμφωνο Σταθερότητα με αυτή την πρόταση. Γιατί η πρόταση της Ντοβίλ ε, αποδυναμώνει όχι μόνο τι προτάσει της Task Force αλλά και το πακέτο της ε, Κομισιόν και δεν το καταλαβαίνω. Το βρίσκω ακατανόητο. Ιδιαίτερα να προέρχεται από τη Γερμανία αυτό. Για δέκα μήνε ζητούσαν πιο αυστηρέ κυρώσει και χτε τι έκαναν, το ακριβώ αντίθετο. Συμφωνούν στην πράξη σε αποδυνάμωση των γενναίων προτάσεων της ε, Κομισιόν. Και ακριβώς τη στιγμή που ο κύριος Τρισέο, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ζητεί πιο γενναίες λύσεις, πιο γενναίες προτάσεις, ακόμα πιο γενναίες και αυστηρές από τις προτάσεις της αρχής προτάσεις της Κομισιόν. Συνεπώς, τι συμπεραίνω εγώ. Έχουμε μία αποστολή εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Να, να αναστρέψουμε την συμφωνία της Ντοβίλ, τη συμφωνία του, το συμβασμό του Καζίνο και να παραμείνουμε προσιλωμένοι στις προτάσεις της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Φερχόφστατ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κον Μπεντήτ για 4,5 λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Ο Γκί δεν μπορεί άλλο να κρατηθεί. Βρήκε ένα κολπάκι και ο Σούλτ ήταν καλός, ναι. Μου επιτρέπετε, έχω κι εγώ μια ιδέα τώρα. Γνωρίζετε όλοι Εκείνο το, την ταινία Ζουλ και Ζιμ. Υπάρχει μια γυναίκα, η κυρία Μέρκελ, ο Ζιμ ξέρουμε ποιο είναι, είναι ο Σαρκό. Το θέμα είναι ποιο είναι ο Τζιμ. Ο Καμερόν ή ο Μπαρόζο. Ε, εδώ είναι το πρόβλημα για την Κομισιόν. Σήμερα πιστεύω πως το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν πρέπει να συνομιλήσουν ειλικρινά γιατί σήμερα το Συμβούλιο και εκεί είναι το Συμβούλιο και εδώ έχει δίκιο ότι είναι το γαλλογερμανικό δικητήριο έχουν μια πολιτική που δεν είναι κοινοτική. Είναι μια πολιτική που δεν περιλαμβάνει την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πέρα από τις, από τις διαφορές μας που υπάρχουν σήμερα και ο Ζωζεφ Ντόλ έχει δίκιο Σήμερα δικός μας ρόλος είναι να σώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινοτική μέθοδο και για να γίνει αυτό πρέπει η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και εμείς, είτε είμαστε μένει δε, να συνονοηθούμε. να καταλάβουμε ότι σε αυτό το παιχνίδι κανείς δεν θα κερδίσει αν δεν βρούμε μια κοινή γραμμή ανάμεσα σε εμά και στην και στην Κομισιόν και τούμπαλιν. Κύριε Μπαρόζο, σας πιστεύω. Θέλετε φόρο για τις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Εντάξει, σας πιστεύω. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Πώς θα το καταφέρουμε είναι. Δεν αρκεί να λέμε θέλω. Αυτό τα λέει ο γιος μου. Όταν είναι τεσσάρων χρονών λέει θέλω. Το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο αυτό. Πιστεύω πως η Κομισιόν οφείλει όχι να ζητεί όπως το περιβαλλοντικό συμβάλλον το ζήτησε μια νιωστή ε, μελέτη για να δούμε αν όντω είναι τέτοια υποβάθμιση του περιβάλλοντος ώστε να πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που έκανε χθες προχθές για να ζητήσει ακόμα μια μελέτη. Μα έχουμε ένα σωρό μελέτες. Σημαντική μελέτη για τις ε, οικονομικές συναλλαγές και φόρος επ' αυτών θα έδινε στην Ευρώπη 0,01% φόρο. Σημαίνει 80 δισεκατομμύρια ευρώ κάτι τέτοιο. Αν δώσουμε 30 δις μείωση στην ε, εθνική συνεισφορά, δηλαδή μείωση για τους εθνικούς προπολογισμούς, μας μένουν 50 δις επιπλέον για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Με 120 δις μείον 30 κάνει 80, ε, συν 50 κάνει 140. Δηλαδή η απαραίτητη κοινωνική πολιτική μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνα. Και μπορούμε όλες αυτές τις απαραίτητες πολιτικές να τις εφαρμόσουμε. Κερδίζουν και τα κράτη και η Ευρώπη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τα βλέπουμε από ευρωπαϊκή οπτική γωνία τα πράγματα. Και έπειτα κύριε Μπαρόζο, σας ζητάω και, για το, και από το Κοινοβούλιο για τα έλλειμμα. Υπάρχουν διαφόρων ειδών ελλείμματα. Είναι όπως και η χολυστερίνη. Υπάρχει <laughs> ένα θετικό δείκτη και ένα αρνητικό δείκτη. Ένα έλλειμμα το οποίο επενδύει και άρα δίνει προοπτικές σε μια χώρα και στην Ευρώπη, αυτό δεν είναι αρνητικό έλλειμμα. Αν όμως επενδύουμε όπως το κάνουμε στις ε, χτεσινές ε, βιομηχανίες που δεν είναι παραγωγικές, μιλώ για τον άνθρακα, όπου επενδύουμε κάτι το οποίο είναι στην ουσία να καταστρέφουμε χρήματα γιατί δεν συγχρησιμεύει σε τίποτα, χάνουμε. Αν όμω επενδύσουμε στι αυριανέ ε, ενέργειε και στι αυριανέ παραγωγές, κερδίζουμε. Άρα λοιπόν αυτό που οφείλουμε να κάνουμε και εδώ, το αυτό το ζητώ και από του φιλελεύθερου. Δηλαδή δεν αρκεί να πούμε σταθερότητα και σταθερότητα μόνο, να φωνάζουμε, αλλά ναι, θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε σε αυτά που πρέπει να κάνουμε και σε αυτά που δεν πρέπει πλέον να κάνουμε. Να μην λέμε μόνο έλλειμμα, αλλά να λέμε ότι αυτό δεν είναι παραγωγικό, ενώ αυτό αντίθετα είναι. Αν συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτά, θα είναι δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να αντισταθούμε στους μόνιμους στη μόνιμη χειραγώγηση του Συμβουλίου. Σήμερα το πρόβλημα είναι ότι πολλές κυβερνήσεις θέλουν να μειώσουν την ευρωπαϊκή πολιτική διάσταση. Και δικός μας ρόλος είναι να υπερασπιστούμε και να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική διάσταση, διότι αν αυτής δεν θα τα καταφέρουμε. Βλέπετε κύριε Μπαρόζο, έχουμε κοινό συμφέρον, αλλά πρέπει να το τραβήξουμε μέχρι τέλος. Να μην ε, ε, να μην βάζετε τρικλοποδία στο Κοινοβούλιο, αλλά στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Το πως είδατε ήμουνα κάπως ε, τσιλαστικός για το χρόνο γιατί οι παρεμβάσεις σας εξάλλου ήταν πολύ χαριτωμένες εκτός από έντονες. Μιλήσατε για το... τη χολυστερόνη. Νομίζω ότι πραγματικά όλοι σας συμπάθησαν με αυτή την παρέμβαση. Επόμενη παρέμβαση ο κύριος Καμίσκι. Ευχαριστώ. Ακούμε διάφορα αστεία σήμερα, ιστοριούλες. Ε, ακούγοντας ε, τη συζήτηση αυτή σκέφτομαι και την ιστορία. Εγώ πέρασα 18 χρόνια της ε, ζωής μου σε ένα σοσιαλιστικό σύστημα και το ένα συνέδριο του κόμματος μετά το άλλο έβγαζε νέους στόχους και άκουγαν σε όλες αυτές τις χώρες οι λαοί από το κόμμα το πώς θα γίνει η κατάσταση καλύτερη. Εμείς είχαμε Υπουργείο Εσωτερικού Εμπορίου στη χώρα μου, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αντικείμενο. Ακούγοντας λοιπόν τις σημερινές ομιλίες, έχω την εντύπωση πως οι προτάσεις που ακούσαμε από την Κομισιόν είναι μια πρόταση η οποία είναι σχεδιασμένη για να δοθεί στην οικονομική πολιτική, να δοθούν στην οικονομική πολιτική τα πρωτεία έναντι της πολιτικής, γιατί η πολιτική με ομικρογιώτα στα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή κατηγορούν την Ευρώπη και λένε πως ε, η Ευρώπη είναι μια κακή ιδέα, γίνονται λάθη και τα λοιπά και η Ευρώπη είναι ο αποδιοπομπαίος τράβος για τα λάθη των πολιτικών των κρατών μελών. Γνωρίζουν όμως τα κράτη-μέλη πως ε, εάν αποτύχει η οικονομική πολιτική τους θα χάσουμε όλοι. Εγώ βλέπω έναν κίνδυνο στη γαλλογερμανική πρόταση. Θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση στην οποία η καημένη Ελλάδα επειδή είναι μικρή θα παίζει με τους κανόνες αλλά εάν μια χώρα είναι αρκετά μεγάλη θα μπορεί να κάνει τον ταΐ και να ξεφεύγει από τους κανόνες και να τους παραβιάζει. Οπότε χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζω πως ο κύριος ε, Μπαρόζο είναι θέμα θεματοφύλακας της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης και εκτιμώ αυτό το οποίο κάνατε για την ε, Ρώσο-Πολωνική Συμφωνία του Αερίου. Χαίρομαι που λειτουργεί η κοινοτική αλληλεγγύη και υποφελείται από αυτό η Πολωνία. Αλλά θα ήθελα να πω εδώ πέρα κύριε Πρόεδρε πως δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τα γεγονότα. Εάν οδηγηθούμε σε μια κατάσταση στην οποία η καθημερινή πολιτική και ο λαϊκισμός υπερισχύουν τις οικονομικές σκέψεις, τότε μπορούμε να ξεχάσουμε την εμβάθυνση της αγοράς, κάτι το οποίο είναι μια καλή ιδέα. Εμείς ως ε, ευρωβουλευτές γνωρίζουμε πόσο πρέπει να προχωρήσουμε στην εσωτερική αγορά κάθε φορά που λαμβάνουμε λογαριασμό με περιαγωγή για τα κινητά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Ευχαριστούμε κύριε Καμίνσκι. λέει... Το λόγο έχει ο κύριος Λεγιαρίκ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ αν κατάλαβα καλά τον πρόεδρο Μπαρόζο, ξεκινάμε από μια ανάλυση τελείως αντίθετη, γιατί είπατε πως η κρίση έχει πια περάσει, ενώ η Γκουε θεωρεί πως ε, επιδεινώνεται η κρίση. Για να την λύσουμε, εσείς προβλέπετε τη λιτότητα με το Σύμφωνο Σταθερότητας, διατηρώντας την ενίσχυση των κυρώσεων Εμεί πιστεύουμε πω είναι το αντίθετο που πρέπει να γίνει με τη βελτίωση των αμοιβών για την εργασία, μια νέα ε, φορολογία θετική για κάτι τέτοιο και τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, βελτίωση της κοινωνικής προστασίας, υπεράσπιση του δημόσιου τομέα και σοβαρή πολιτική για την απασχόληση. Φοβούμε πω η στρατηγική σα οδηγεί την Ευρώπη να χτυπήσει το κεφάλι τη στον τοίχο. Δεν ακούτε την ένταση των λαϊκών ε, διαμαρτυριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση. Έκτη μέρα χτες εκατομμύρια άνθρωποι διαδήλωσαν στην Γαλλία και τους υποστήριξε το 70% του πληθυσμού. Δεν βλέπετε τον κίνδυνο που μας απειλεί σήμερα. Η ευρωπαϊκή ιδέα που βασίζεται στον ανταγωνισμό, στον ελεύθερο, απόλυτο, στις απόλυτα ελεύθερες συναλλαγές θα σπάσει το κεφάλι της στον τοίχο μέσα στην οικονομική, στον οικονομικό και νομισματικό πόλεμο. Γιατί να μελετήσουμε ένα νέο σύστημα, ένα ταμείο ανάπτυξη ανάπτυξης, ανθρώπινης ανάπτυξης ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μέσω της νομισματικής δημιουργίας θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το χρέος των κρατών και ε, τις εθνικές τράπεζες με βάση ε, επιτόκια που θα είναι ευνοϊκά για, με βάση κοινωνικά κριτήρια. Νέα νομισματική παγκόσμια τάξη αρχίζοντας στηριζόμενη στην κινέζικη πρόταση ενός κοινού ε, νομίσματος συναλλαγών για τις παγκόσμιες συναλλαγές. Όπως έχει κάνει η Βραζιλία και η Ταϊλάνδη, γιατί να μην φορολογήσουμε τα νομίσματα για να περιορίσουμε τις νομισματικές εντάσεις. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής και εκπρόσωπε του Συμβουλίου, νομίζω πως πρέπει να φανταστούμε πια νέε πρωτοβουλίε και να ακούσουμε τους λαού. Σα ευχαριστώ κύριε Λεγιαρίκ. Το, το λόγο έχει ο κύριος Φάρατζ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπαρόζο, οπωσδήποτε εδώ πέρα εξασκείτε την ισχύ που σας έχει δώσει η συνθήκη της Λισαβόνας και κάνετε οτιδήποτε μπορείτε στην παγκόσμια σκηνή και εντός, και εντός Ένωσης για να αποκτήσετε όλες οι ιδιότητες του κράτους και πουθενά και βεβαίω αυτό καθίστε πιο προφανέ με το να θέλετε να επιβάλλετε άμεσο φόρο στου λαού αυτή τη Ευρώπη. Βεβαίω, τον παλιό καιρό υπήρχε, υπήρξε ένα πολύ επιτυχημένο κίνημα ανεξαρτησίας με σύνθημα καμία φορολογία χωρί εκπροσώπηση. Και εσεί οπωσδήποτε δεν είστε εκπρόσωπο, δεν σα ψήφισε κανεί και δεν μπορεί να σα απομακρύνει. Οπότε νομίζω πω κάνετε λάθο με αυτό τον φόρο. Και τι ακριβό κλαμπ έχει γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από δύο χρόνια η Βρετανία έδινε 3 δισεκατομμύρια λίρε του χρόνου. Φέτος ήταν 6 δισεκατομμύρια, του χρόνου θα είναι 8 δισεκατομμύρια λίρε. και μετά 10 δισεκατομμύρια λίρε. Και τώρα ακούμε πω θέλετε να ανακαλέσετε τη Βρετανική επιστροφή που σημαίνει πως μέχρι το 2013 η συνεισφορά μας θα είναι 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα έχει τετραπλασιαστεί μέσα σε 6 χρόνια. Και βεβαίως όταν το δουν και το αντιληφθούν αυτό οι ε, Βρετανοί φορολογούμενοι θα πούν πως δεν μπορούμε να πληρώσουμε πλέον αυτή την πολυτέλεια που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό το οποίο έκαναν στην Ντοβίλ Σαρκοζή και Μέρκελ, αυτό το οποίο φοβάστε, εγώ ελπίζω να συμβεί. Να έχουμε μια νέα συνθήκη και εσείς φαίνεται πως την υποστηρίζετε και να τεθεί σε δημοψήφισμα σε πολλές χώρες, ειδικά στη Βρετανία και θα συμπεράνει ο Βρετανικός λαός πως είναι πάρα πολύ κακή συμφωνία για την Βρετανία. Θα ψηφίσουν να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, ναι, εμείς θέλουμε να φύγουμε. Ευχαριστώ. Κύριε κύριο Σούλτ, μια ερώτηση προ τον κύριο Φάρατ θέλει να θέσει. Κύριε Φάρατ, έχω ένα ερώτημα. Ίσως μπορείτε να μας το απαντήσετε. Ανισχύετε τόσο πολύ για τη Βρετανικό Ταμείο. Όπως και εσείς έτσι και εγώ είχα την δυνατότητα να επιλέξω στην αρχή της θητείας μου από πού θα πληρώνω, από το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ήθελατε να μας πείτε εάν επιλέξατε να πληρώνεστε από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από το Εθνικό Σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας. Πρέπει να καταργηθεί νομίζω αυτή η ιδέα των ευρωπαϊκών χρημάτων αν δεν υπάρχει άμεσος φόρος, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι δικά μας τα λεφτά. Πληρώνουμε πάρα πολύ, είμαστε καθαρός εισφορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουμε κανένα απολύτως οικονομικό όφελος. Δικά μας είναι τα λεφτά. Πρόεδρε Μπαρόζο. No, ε, Συνήθω δεν παρεμβαίνω, αλλά υπάρχει ένα διαδικαστικό ζήτημα που θα ήθελα να θίξω. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριο Φάρατζ. Ε, αναφέρεται σε μένα λέγοντα δεν έχετε εκλεγεί. Ασφαλώς δεν έχω εκλεγεί από εσά. Έχω εκλεγεί όμω από το κοινοβούλιο, από αυτό το κοινοβούλιο. Εξελέγει μέσω μυστική πληροφορία από αυτό εδώ το κοινοβούλιο. Και εσεί ανήκετε σε αυτό το κοινοβούλιο. Οπότε αποτελεί έλλειψη σεβασμού προς, το, προς την Κομισιόν αλλά και προς το Κοινοβούλιο να λέτε ότι εγώ και τα μέλη της Κομισιόν δεν έχουμε εκλεγεί. Ωραία. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εγώ δέχομαι τα όσα είπε ο Πρόεδρος Μπαρόζο. Νομίζω πως είναι σωστά τα όσα είπε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σόζα Βάγκνερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να δω μπας και καταφέρω να ηρεμήσω αυτή την ε, πολύ ζωντανή συζήτηση. Είναι κρίμα που εξακολουθούν μαζί με την Ευρωπαϊκή στο G20, να βρίσκονται και κάποιες ε, χώρες ε, που δεν θα έπρεπε. Ε, είναι μια ανομαλία που αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ε, κόσμο. Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε μια κοινή θέση σε αυτό το Παγκόσμιο Φόρουμ. Και ποια θα ήταν αυτή η κοινή θέση. Ταπεινά πιστεύω ότι δεν, πρώτον δεν πρέπει να καθυστερήσουμε την υιοθέτηση μιας παγκόσμιας συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κρίσης. Όχι μόνο οικονομικής όμως συμφωνίας. Δεύτερον, η Ευρώπη θα πρέπει να διατηρήσει το ευρώ ως ε, νόμισμα αναφοράς. Αν θέλετε ως άγκυρα για να αποφύγουμε η ε, αναστάτωση στην αγορά μας ε, οδηγήσει να επαναλάβουμε τα λάθη που κάναμε. Τρίτον, το ευρώ θα πρέπει να αποτελεί, να σηματοδοτεί μάλλον τις δημοκρατικές αρχές και τι ε, ελευθερίε που προωθεί και προασπίζει η Ευρώπη στον κόσμο. Στον, ε, στην, στον παγκοσμιοποιημένο μα κόσμο χάνει αυτό ο οποίο ε, παίζει μόνο τα εθνικά χαρτιά του. Σα ευχαριστώ κύριε Σόσα Βάγνερ. Το λόγο έχει ο κύριο Κάρα για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση καταδεικνύει ένα πράγμα πως η συμφωνία της Ντοβίλ μας εμποδίζει να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Είναι βήμα προς τα πίσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας δείχνει πως ο κύριος και η κυρία δεν έχουν μάθει τίποτα από το 2005 όταν ξεκίνησαν να υποβαθμίζουν το σύμφωνο σταθερότητα. Πρέπει να ξεπεράσουμε το 2005. Πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση στους εθνικισμούς και στα, στο διάφορα μηχανισμούς που μπλοκάρουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αυτό το κάνουμε με την έκθεση ΦΕΙΟ και με την καθημερινή μας νομοθετική εργασία. Σε αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθούμε και να μην μας εμποδίζουν σε αυτό. Ούτε εδώ μέσα σε αυτή τη συζήτηση πρέπει να αναζητήσουμε την ε, λύση και νομίζω πως η έκθεση αυτή των τεσσάρων αυτών ομάδων λέει πάρα πολλά πράγματα. Η δημοσιονομική πολιτική δεν αποτελεί πολιτική μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα γίνει η μείωση των ελλημάτων, η οποία όμως δεν μπορεί να γίνει με τη μηχανή του γκαζόν. Πρέπει να γίνουν και επενδύσεις. Η έκθεση αυτή εδώ πέρα λοιπόν δίνει μια σαφή απάντηση. Θέμε περισσότερη Ευρώπη ως μέρος της λύσης. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε μία ένωση κοινωνική, μία ένωση η οποία θα έχει χαρακτηριστικά που θα ευνοούν όλους τους πολίτες από κοινού. Λοιπόν θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Task Force και η μέθοδος Ντοβίλ έχουν αποτύχει. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Στίβεν Χιούς για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, η Task Force ε, υπέβαλε την έκθεσή της ε, με προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης και δημοσιονομική πειθαρχία. Όμως αυτό είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητας και πρόκειται μόνο για προτάσεις. Είμαι σίγουρο ότι οι Υπουργοί ΕΚΟΦΗΝ ε, θα ήθελα να τελειώσει και αυτή η διαδικασία, αλλά δυστυχώ είναι η αφετηρία. Βρισκόμαστε στην αφετηρία της νομοθετικής διαδικασίας και ελπίζω ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα αντιληφθούν ότι το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να γίνει σε, πλαίσιο, σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σε συνεργασία με το Συμβούλιο. Ε, θέλουμε να γίνει ένα άλμα στην αποτελεσματικότητα της οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά η προτάσεις ε, αποτελούν οπισθοδρόμηση ό,τι αφορά την ευημερία στην Ευρώπη. Οι προτάσεις ε, ενισχύουν τα όργανα τα οποία εστιάζονται στη δημοσιονομική πειθαρχία και μόνον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, η Οικονομική Ένωση δεν θα επιτευχθεί αν δεν εξασφαλίσουμε την ισορροπία διότι με τις προτάσεις αυτές θα διαστραφούν οι οικονομικές πολιτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο ως μακροοικονομικές πολιτικές εις βάρος της απασχόλησης των, της ανάπτυξης των επενδύσεων. Δεν χρειαζόμαστε άλλη μια task force. Χρειαζόμαστε η Κομισιόν να χρησιμοποιήσει τις, το δικαίωμα πρωτοβουλία της για να υποβάλει προτάσεις που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της επενδύσεις και την ε, απασχόληση. Το Κοινοβούλιο ε, έχει τεράστια ευθύνη στους επόμενους μήνες από τη δική του μεριά. Πρέπει να κάνουμε μερικές αλλαγές στην έκθεση ΦΕΙΟ ε, πριν την υιοθετήσουμε. Τρεις βασικές αλλαγές. Πρώτον, να αντιμετωπίσουμε το θέμα των σημαντικών ανισορροπιών ε, να ληφθούν υπόψη πολύ περισσότερο οι δείκτες ε, ανεργίας. Μετά έχουμε την ποιοτική αξιολόγηση των δημόσιων χρεών και, τους, και, και οι μηχανισμοί ε, αντιμετώπισης των, των υπερβολικών χρεών θα πρέπει ε, να λαμβάνουν υπόψη περισσότερα κριτήρια. Ε, μετά για την οικονομική διακυβέρνηση δύο θέματα, δύο σχόλια. Το Συμβούλιο θα πρέπει να αναλάβει την τελική πολιτική ευθύνη και να, και να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία όχι μόνο το κοφίνα αλλά και τα υπόλοιπα συμβούλια. Τέλο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίση να συμμετάσχει πλήρω στη διαδικασία για να εξασφαλίσουμε τον υψηλότερο βαθμό ε, δημοκρατική νομιμοποίηση. Το ευρωπαϊκό, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι πολύ μειωμένος για παράδειγμα. Θα πρέπει να ε, υποβάλουμε προτάσεις για ενίσχυση της συμμετοχής του Κοινοβουλίου. Έχουμε ήδη υποβάλει αυτές τις προτάσεις εμείς και ελπίζω ότι θα τις ε, δεχτούν και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. E ευχαριστώ κύριο Σμιτ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι. Το τελευταίο έτος είδαμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λάβει σημαντικές αποφάσεις όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Τις τελευταίες μέρες όμως είχαμε κάποια απογοήτευση όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πιο αυστηρές γραμμές προπολογισμού, διστάζουν η Γαλλία και η Γερμανία. Και εμείς λέμε μην πειράξετε την πρόταση του Όλη Ρεν. Τελεία. Ε, επίσης πρέπει να ευχαριστήσω την ε, κύρια Μπερές ε, και την ψηφοφορία στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων που δείχνουν πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε. Μια τροπολογία που έχουμε να κάνουμε είναι πως ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πρέπει να επιβληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να οδηγηθούμε ξανά σε εθνικισμούς στην Ευρώπη. Έχουμε μια οικονομία που ασύζεται στην αγορά, ξεκάθαρο πλαίσιο, ελεύθερο εμπόριο που δημιουργεί πλούτο και ευημερία. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο ενωμένη, πιο ισχυρή Ευρώπη. Πολύ απλά χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Οι δυνατότητες κυρώσεων που προτείνονται στην αρχή μιλούσαν μόνο για τις χώρες του ευρώ. Εδώ πέρα λοιπόν θα θέλαμε να αλλάξει διατύπωση για να συμπεριλάβουν και τις 27 χώρες και θα καταθέσουμε μια σχετική τροπολογία που ελπίζω να την στηρίξετε. Η δε η συγγήτρια των σοσιαλιστών λέει πως θα το κάνει. Στα αγγλικά λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν στο μέγιστο όλες τις προτάσεις οικονομικής διακυβέρνησης αναγνωρίζοντας πως για μέτρα εκτός Ευρωζώνης αυτό θα γίνει σε εθελοντική βάση. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να οδηγηθούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που κινδυνεύει να διαλυθεί. Ευχαριστώ συνάδελφε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Καμφέν για δύο λεπτά. Ναι, κύριε Μπαρόζο και κύριε Ρεν, πραγματικά ελπίζω ότι θα δείτε τα όσα έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα, έκθεση Μπερές και Φέγιο, γιατί φυσικά είμαστε σε ένα πλαίσιο συνομοθε... Ε, για την οικονομική διακυβέρνηση και ειλικρινά μπορώ να σας πω ότι κάναμε τουλάχιστον με τις τέσσερις πολιτικές ομάδες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι υπέρ της Ευρώπης έχουμε κάνει προσπάθειες για συμβαστικές λύσεις πολύ δυναμικές και τελειώνει αυτή η συζήτηση μιλάμε από τη μια μεριά μιλάμε για το προπολογισμό μετά μιλάμε για φορολόγηση, μετά μιλάμε για διακυβέρνηση κτλ. Η αλήθεια είναι πως εδώ είναι δικό σας ρόλος να το κάνετε αυτό ε, και εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε να προτείνουμε ένα σφαιρικό, ένα γενικό πακέτο μέσα στο πλαίσιο της έκθεσης Μόντι. Ε, το ίδιο προσπαθεί να κάνει και ο Μισελ Μπαρνιέ στην εσωτερική αγορά. Εγώ περιμένω το πακέτο του Μπαρόζο να που θα πει να, έτσι θα βγούμε από την κρίση. Όχι μόνο για τη μακροοικονομική διακυβέρνηση, αλλά πώ θα συνδέσουμε τρία-τέσσερα μακροοικονομικά ντοσιέ ε, φορολογία, προϋπολογισμός, μακροοικονομία. Αν το κάνετε αυτό θα, θα δείτε μεγάλη πλειοψηφία να σας στηρίζει στο Κοινοβούλιο. Γιατί αν μείνουμε ας πούμε μόνο στο θέμα των, ε, της δημόσιας οικονομίας. Εσείς οι ίδιοι στην υπηρεσία σας λέγατε πριν από τρία χρόνια ότι η Ισπανία ήταν αυτή που σεβόταν καλύτερα το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το, η κρατική οικονομία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Και τώρα η Ισπανία το πρόβλημα ήταν ότι η ανατραχή προήρθε από αλλού και βρίσκεται σε μια φρικτή κατάσταση. Το ίδιο και η Ιρλανδία. Και ε, στις διάφορες εκθέσεις, τα όσα σας παρουσιάσαμε σήμερα και αύριο, Ακριβώς περί αυτού πρόκειται, η, προ... η ισόρευση αυτών των προβληματικών. Ναι, πρέπει να ενισχυθεί η δημοσιονομική λιτότητα, βεβαίως, αλλά για να μην μεταφραστεί αυτό από, σε κοινωνικέ διατραχέ και δηλαδή μόνο περικοπέ στι δημόσιε δαπάνε, θα πρέπει να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πακέτο για να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσει και για ένα φορολογικό πακέτο για να μπορέσουν τα κράτη να συλλέξουν κάποιου φόρου. Τελευταία ερώτηση κύριε Μπαρόζο. Είστε πραγματικά υπέρ ή στηρίζετε πραγματικά το θέμα της ε, παγιωμένης φορολογικής ε, βάση. Ε, δέκα χρόνια είναι στα συρτάρια τη Κομισιόν, δέκα χρόνια το εμποδίζετε. Κάντε το τώρα επιτέλους. Σα ευχαριστώ. Τώρα έχει το λόγο ο κύριο Ρόμπερτ Ζιλ για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε της Επιτροπής από τη συνάλφη. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το, τους εισηγητές και τους ε, διότι έχουμε καταλήξει σε, μια, σε ένα συμβασμό. Δύο μόνο θέσεις ε, θα ήθελα να σχολιάσω μετά από διαμεθοριακές επενδύσεις σε διάφορα κράτη-μέλη μετά το 2004 αυξήθηκαν τα ιδιωτικά χρέη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων μάλιστα δέκα πλασιάστηκαν, δέκα πλασιάστηκαν. Επίσης υπάρχουν και συναλλαγματικοί κίνδυνοι για αυτούς που έλαβαν τέτοιου είδους ε, διαμεθοριακά δάνεια ε, διασυνοριακά δάνεια να το πούμε καλύτερα ταυτόχρονα για δημοσιονομικούς λόγους αυξάνονται οι φόροι, οπότε τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν ξέρουν πώς θα επιστρέψουν τα δάνεια αυτά, τις πιστώσεις. Αυτό δεν αναφέρεται πολύ σαφώς στην έκθεση αυτό το πρόβλημα. Δεύτερο, σε σχέση και πάλι με το πρώτο, στα νέα κράτη-μέλη που το ΑΕΠ ε, έχει πέσει σε επίπεδο που, στο επίπεδο που βρισκόταν πριν την ένταξή του το 2004. Έχουμε τα, ταυτόχρονα τα ιδιωτικά δάνεια που έχουν δεκαπλασιαστεί, το δημόσιο χρέο, το οποίο επίση έχει πενταπλασιαστεί. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα δημιουργούνται ε, με την πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι δηλώσεις της Γερμανίας και της Γαλλίας, ε, η αποκαλούμενη συμφωνία του Ισντοβίλ είναι απαράδεκτες και, και αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο αυτών που δίνουν τις ε, ε, διαταγές. Αποκαλύπτει την ανυπομονησία, την υπεροψία και την επιθετικότητα απέναντι στους εργαζόμενους και μέσω των προτάσεων και των φιλελεύθερων αυτών πολιτικών και των αντικοινωνικών ε, πολιτικών. Πολιτική ανταγωνισμού στην Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία που προβλέπονται ήδη μια γενική απεργία για τις 24 Νοεμβρίου. Οι υπεύθυνοι της ε, ηθήνοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγνωρίσουν την αποτυχία αυτών των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που αυξάνουν την ε, ενεργεία της κοινωνικές ανισότητας, την φτώχεια και προκαλούν ύφεση στις χώρες που έχουν πιο αδύναμες οικονομίες όπου οι κοινοτικοί φόροι μπορεί να προκαλέσουν μια πραγματική κοινωνική καταστροφή. Αυτό συμβαίνει. Πού είναι εκείνες οι υποσχέσεις που δόθηκαν για τη φορολογία των οικονομικών συναλλαγών για την απαγόρευση των κερδοσκοπικών προϊόντων. Διαμαρτυρόμαστε. Διαμαρτυρόμαστε με πολλά εκατομμύρια ανθρώπων, εργαζόμενων που απειλούνται από τη φτώχεια και από διάφορες μορφές ε, μιζέρια. Οι νέοι κινδυνεύουν και τα παιδιά από τη φτώχεια. Ποια μέλλον αξιοπρεπές θα έχουν σε μια τέτοια φάση. Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να πάψουν για να έχουμε μια πραγματική κοινωνική Ευρώπη, μια Ευρώπη προόδου και ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους που έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν να τερούν αυστηρά το χρόνο τους γιατί διαφορετικά θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία ψηφοφορίας πολύ αργά. Προβλέπονται πολύ πολύ χρονοβόρες ψηφοφορίες. Λοιπόν, θα σας παίρνω το λόγο άμα ξεπερνάτε το χρόνο σας. Και τώρα ο κύριος Ιμπράζας για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω δύο λόγια για τις εργασίες της Ειδικής Επιτροπής ε, για την ε, κρίση. Ε, το έργο της ήταν πολύ καλό και οι προτάσεις επίσης. Το ιδανικό θα ήταν όλες αυτές οι προτάσεις της Επιτροπής να ενταχθούν στις προτάσεις Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν θα πρέπει να γνωρίσει το πιο βασικό. Χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό ρυθμίσης και εποπτείας για όλες τις χρηματοοικονομικές αγορές, για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα και όλα τα, και όλους τους φορείς αυτού του τομέως. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά της ε, ανεργίας ε, ε, που θα ενταχθούν στον αγώνα εναντίον της στόχιας. Ε, το, θα πρέπει να εστιαστούμε ιδιαίτερο στην απασχόληση των νέων. Θα πρέπει να λάβουμε επίσης στην αποφάσεις σχετικά με τις ε, επενδύσεις υποδομές, της, ε, τον τομέα των μεταφορών, της στέγασης και της ενέργειας. Το τέλειο θα ήταν ε, ένα χρόνο μετά η Κομισιόν να μπορούσε να πει ε, ότι αυτά που προτείναμε δεν έμειναν κενό γράμμα και ότι υλοποιήθηκαν με κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που τηρήσατε το χρόνο. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Κριστίνα Μορβάη για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δις συζήτησε το θέμα της στόχες ήδη. Και γι' αυτό και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουν λύπη στους ότι η κατάσταση των Ευρωπαίων επιδεινώνεται. Αυξάνεται η ανεργία, η... φτωχοί πολλαπλασιάζονται. Συνήθως αυτό γίνεται μετά από μια φυσική καταστροφή, ένα τσουνάμι, όμως όχι. Αυτά είναι όλα συνέπειες των αποφάσεων των Ευρωπαίων Ιθινόντων ε, και προέρχονται, οφείλονται μάλλον στην νεοφιλελεύθερη πολιτική που ε, εσείς ακολουθείτε. Αυτή τάσει επιδεινώνουν τη φτώχεια, συνεχίζεται η ταλαιπωρία και αν δεν αλλάξετε πορεία, αν δεν ακολουθήσετε άλλες αρχές δεν θα έχουμε καλό τέλος. Είναι όπως όταν ένας γιατρός βλέπει πως δεν θεραπεύεται ο άρρωστος και ως αγωγή συνεχίζει να του προτείνει την ίδια αγωγή, την φαρμακευτική, με πιο αυστηρό έλεγχο, τιμωρώντας τον ασθενή αν αυτός ε, δεν πάρει το φάρμακό του. Εδώ πρόκειται για ένα, μια επιλογή μια επιλογή που ανάμεσα στα διάφορα συστήματα αξιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν έθετε το ερώτημα ποια είναι η καλύτερη απόφαση από την άποψη του κέρδους, του χρήματος του και του ωφέλους των πολυεθνικών και των τραπεζών. Και ποτέ δεν αναζήτησε την καλή λύση υπέρ των ε, απλών ανθρώπων. Χρειάζεται ο ανταγωνισμό, αλλά θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη. Από εδώ και μπρο θα πρέπει να λεφθούν οι σωστέ αποφάσει. Σα ευχαριστώ. κυρία Βόρτμαν Κόλ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν θετικά μηνύματα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνο να επιδεινωθεί η κρίση. Το τραπεζικό σύστημα δεν είναι ακόμα σταθερό και για αρκετά κράτη-μέλη απειλούν οι περικοπές να τα ελλείμματα να ξεφύγουν εάν δεν κάνουμε περικοπές. Κύριε Πρόεδρε, τα αποτελέσματα της ε, Task Force ε, είναι γνωστά, αλλά βεβαίως, ε, όπως είπε ο κύριος Επέτροπος, μπορούμε ακόμα να εργαστούμε γρήγορα, αλλά βεβαίως με βάση τις προτάσεις της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι το Συμβούλιο διατεθειμένο να αποδεχθεί κάτι τέτοιο. Επίσης δεν θα πρέπει να αλλάξει αυτή τη στιγμή η συνθήκη, αλλά θα πρέπει να ληφθούν γρήγορα κάποια μέτρα για να κάνουμε αυτά το οποίο είναι αναγκαίο και δυνατόν εντός της συνθήκης της Λισαβόνας και αυτό το κοινοβούλιο τώρα έχει να παίξει ένα ρόλο ως συνομοθέτης και μέσω του Συμφώνου Σταθερότητας και θα πρέπει να το κάνουμε αυτό για να έχουμε μια στιβαρή οικονομική ένωση με ένα στιβαρό Σύμφωνο Σταθερότητας και ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ κυρία Βόρτμαν. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σέρτζιο Κομφεράτη για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολύ βαριές για την ε, κοινωνία όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Αν δούμε την κοινωνική πτυχή, φτάνουμε γρήγορα στο συμπέρασμα ότι εξάλλου έχει προσανατολίσει πολλές από τις εργασίες της Κομισιόν και μάλιστα ότι τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμα. Η ανεργία θα αυξηθεί και τα ισχνά σημεία ανάκαμψης που φαίνονται σε διάφορες χώρες δεν αρκούν για να εγγυηθούν τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως θα είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε την πιο οξία φάση από κοινωνική αυτή άποψης αυτής της κρίσης που δημιουργήθηκε από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και γρήγορα έπληξε το οικονομικό και το κοινωνικό ε, σύστημα. Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να Έχουμε στη διάθεσή μας επιπλέον μέσα άμυνας για τα άτομα τα οποία πλήττονται περισσότερο. Μια υπόθεση οδηγίας πλαισίου για το μίνιμουμ ε, εισόδημα, εγγυημένο εισόδημα όλων των Ευρωπαίων για να, αντιστα... τη φτώχεια αλλά και για να προβλέψουμε αυτούς που τους επόμενους μήνες θα ε, χτυπηθούν ανελέητα από την κρίση. Από την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρξει και ανάκαμψη, ε, ανάπτυξη, η οποία χρειάζεται επενδύσεις ε, στοχευμένες. Ε, θα πρέπει να διοχετευθεί ένα σημαντικό τμήμα των, διαθέσιμων πόρων. Το προπολογισμό της Ένωσης δεν αρκεί και γι' αυτό και η Κομισιόν σαφώς υπέδειξε την απέτηση για επιπλέον πόρους που θα πρέπει να δαπανηθούν για επενδύσεις σε υποδομές αλλά και ε, που θα καταναλωθούν για την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ε, μιλάμε για ευρωομόλογα αλλά και για τη φορολόγηση των οικονομικών συναλλαγών. Δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικέ λύσεις. Ελπίζω πως το Κοινοβούλιο αυτό θα το ε, επιβεβαιώσει καθώς και η Κομισιόν θα το επιβεβαιώσει. Ευχαριστούμε κύριε Κοφεράτη, ο κύριος Κλίντς για 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην ε, κορύφωση της κρίσης οι χώρες των G20 υποσχέθηκαν να αντιμετωπίσουν Κίνα την από κοινού τη αθεροποίηση των χρηματαγορών. Δεν υπάρχουν όμως σήμερα ακόμα κοινέ ε, απαντήσεις. Τα δε μέτρα που ελήφθησαν ήταν σε μεγάλο βαθμό εθνικά. Το δε πνεύμα που επικρατούσε έχει φύγει και έχουμε ε, περάσει ξανά στο business as usual. Ο Δε Marvin King της Τράπεζας της ε, Αγγλίας λέει πως δεν έχει ακόμα υπάρξει ανάγκη για να δράσουμε προς το συλλογικό συμφέρον. Λοιπόν, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμο. Χρειαζόμαστε η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Πρέπει να δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε τα έργα υποδομής σε ενέργεια και τηλεπικοινωνίες και να δούμε τι θα γίνει με την εσωτερική αγορά εργασία για να επιτύχουμε του στόχου για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Χρειαζόμαστε καινοτόμε πηγές χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε το δυναμικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χρειάζεται περισσότερη κοινοτική και όχι διακυβερνητική μέθοδο. Το να παραμείνουμε στάσιμοι σημαίνει πω πάμε προ τα πίσω και η κρίση στην Ευρώπη δείχνει πως η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη δεν υπάρχουν χωρίς πειθαρχία οι προτάσεις του Επιτρόπου Όλη και του κυρίου Φαν θέλουν βεβαίως να διασφαλίσουν τα, της, τα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δυστυχώς όμως χτες όλα αυτά το γαλλογερμανικό ντουέτο τα πέταξε στα σκουπίδια. Κάτι το οποίο βέβαια απογοητεύει ακόμη μια φορά τους πολίτες. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ε, η κυρία Σουίνμπουρν για ένα λεπτό. Τα θέματα της σημερινής συζήτησης έχουν ένα κοινό παρανομαστή, την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Το πώς θα κάνουμε πιο αποτελεσματική τη διαχείριση του κινδύνου. Διαχείριση του κινδύνου που προέρχεται από τις οικονομικές αγορές, το δημόσιο χρέας ή από τις παγκόσμιες ανισορροπίες. Ε, είτε, προ, είτε αυτοί οι κίνδυνοι προέρχονται από τι τράπεζε είτε από τα Υπουργεία Οικονομικών, θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση με βάση κοινού κανόνε ε, για τη δημοσιονομική πειθαρχία του κρατικού και του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση ότι θα ε, δώσουμε αρκετέ δυνατότητε ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα χρησιμοποιηθούν τα επαρκή ποιοτικά εργαλεία χρηματοοικονομικά εργαλεία, ε, ενώ ταυτόχρονα θα είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα καινούργια χρηματοοικονομικά μέσα. Θα πρέπει επίσης οι προπολογισμοί να καθορίζονται με βάση την πλήρη γνώση των κινδύνων. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, αν υποστηριχθεί από ευρωπαϊκά ομόλογα θα πρέπει πρώτα αυτό το θέμα να συζητηθεί ε, πολύ σοβαρά και αναλυτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Χουντής για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλώντας εκ μέρους της ομάδας της Γκουε για το κείμενο Μπερές, για το κείμενο της κρίσης και δικαιολογώντας γιατί δεν θα την ψηφίσουμε, θέλω να σας πω κύριε Πρόεδρε, επειδή πλεόνασαν οι ιστορικές αναφορές, ότι το σημερινό κείμενο σε σχέση με το αρχικό κείμενο που είχε καταθέσει η συγγήτρια μοιάζει σαν τους παλιούς πάπυρους, σαν τις παλιές περγαμηνές που πάνω στο αρχικό τους γραφεί έξυναν και έγραφαν καινούργια πράγματα ενώ στο κείμενο έμειναν υπολείμματα αυτό που λέγεται παλίμψιστο. λοιπόν από το άγριο ξύσιμο που έγινε στην αρχική τίμια και ειλικρινή προσπάθεια της εισηγήτριας να καταγράψει τις αιτίες της κρίσης και να δώσει τολμηρές προτάσεις ξύσιμο που έγινε από την πλευρά της συμμαχίας των σοσιαλιστών και της ευρωπαϊκής δεξιάς προέκυψε ένα κείμενο όχι πια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου του μόνου δημοκρατικού θεσμού μέσα στο ινστιτούτο της ε, ευρωπαϊκής ένωσης αλλά είναι κείμενο κομισιόν δηλαδή ένα κείμενο που αποκρύβει τις αιτίες της κρίσης και ένα κείμενο που δεσμεύει την πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης στις πρωτοβουλίες μέρκελ σαρκοζή και task force. κάναμε προτάσεις για να βελτιωθεί το κείμενο κριτικάραμε το σύμφωνο σταθερότητας κριτικάραμε τη λειτουργία της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας έχουμε καταθέσει τροπολογίες για να δούμε αν όσοι μιλούν και σήμερα για λαθεμένο δρόμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν εννοούμε το ίδιο πράγμα. η δική μα πρόταση εμπνέεται ε, κύριοι συνάδελφοι από τα κινήματα σήμερα στη γαλλία από τα κινήματα των εργαζομένων στη γερμανία που μειώνονται τα εισοδήματά του για να κάνει δωροδοκίε η siemens από τα κινήματα των εργαζομένων στην ελλάδα που αντιμετωπίζονται σήμερα σαν πειραματόζωα. ένα κείμενο λοιπόν που έχει καταλήξει με τέτοια μορφή δεν μπορούμε να το δεχτούμε. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Μποργέτζο για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να ακούσουμε τις ε, συμβουλές του βραβείου Νόμπελ Μωρίσα Βαλέ που ζητούσε ε, να κλείσουν αυτές οι τράπεζες οι κερδοσκοπικές και οι χρηματοπιστωτικές ε, τέτοιες δράσεις. Και έπειτα, φορολογία των ευρωπαϊκών επενδύσεων. No tax in Europe, άμα περάσει αυτή η πρόταση, μη να ανησυχείτε θα γίνει μαζική διαμαρτυρία. Ο Ευρωπαίος πολίτης δεν θέλει να πληρώνει για μια υπηρεσία που δεν έχει και έχει απόλυτο δίκιο να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τις τράπεζες. Μα τι κάνουν οι τράπεζες μέσα στη full κρίση οικονομική και χρηματοπιστωτική. Αγοράζουν τίτλους που συμπεριλαμβάνουν ένα σωρό σαχλαμάρες, παράγωγα κτλ και, ε, και εμεί τι κάνουμε, αφήνουμε να συνεχίζεται. Είναι η Ευρώπη των τραπεζιτών. είναι προφανέ. Το είπαν και οι αρχηγοί των ε, διαφόρων μασονικών στον Εμεί τι, τι χρειάζεται να κάνουμε, Να αντιμετωπίσουμε τι κερδοσκοπίε με μόνο μία μέθοδο. Δηλαδή, μόνο με τη ε, φορολόγηση των διαπραγματεύσεων. Των διαπραγματεύσεων και μάλιστα σε μετρητά θα πρέπει να πληρώνονται αυτά. Ευχαριστώ. η κυρία Πιετικάινεν για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, δύο χρόνια από το ξέσπασμα της ε, κρίσης και έξι μήνες μόνο έχουν περάσει από την ελληνική κρίση και βλέπουμε πως πλέον δεν υπάρχει καμία διάθεση στα κράτη-μέλη. Σήμερα έχουμε ένα σαφές μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από πέντε ομάδες που στηρίζουν τις εκθέσεις Μπερές και ΦΕΗ. Όπως χρειαζόμαστε πιο συνεκτική οικονομική πολιτική, περισσότερη Ευρώπη, ένα καλύτερο σύμφωνο σταθερότητας και ενίσχυση των μηχανισμών του. Και πραγματικά πρόκειται για χαστούκι στους Ευρωπαίους πολίτες, αυτό το οποίο αποφάσισε δηλαδή πρόσφατα το ε, Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ανάπτυξη οικονομικά υπεύθυνη και σωστή για το περιβάλλον και αηφόρο και καλύτερους μηχανισμούς για την Ευρώπη 2020 και χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση για να υποστηριχθεί αυτή η γραμμή και ε, του φόρου αυτού στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές συμπεριλαμβανομένου κάτι το οποίο άκουσα να υποστηρίζει και η Κομισιόν και δεν και πρέπει να έχουμε βέβαιω πιο ενωμένη ευρωπαϊκή φωνή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καλύτερη ρύθμιση και έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε και χρειαζόμαστε για να καταλήξω μια πρωτοβουλία της Κομισιόν. Η Κομισιόν να δράσει προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών αντί να κάνει μόνο διάφορες task force. Ευχαριστώ. Μπούλμαν για δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, Προεδρία του Συμβουλίου θα μπορούσε αυτή η στιγμή να είναι η στιγμή των μεγάλων απαντήσεων, αλλά δεν το βλέπω. Αυτό το οποίο έχουμε επιτάπητος για τη λεγόμενη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας δεν είναι μεγάλη απάντηση. Είναι και πάλι ο ελάχιστος κοινό παρονομαστή. Είναι το ελάχιστο στο οποίο μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Η Κομισιόν συγχαρητήρια βεβαίως γιατί και εσείς κάθεστε μαζί στο τραπέζι, δεν τα κατάφεραν μόνο τους τα κρατημέλη και συγχαρητήρια βέβαια και στο Συμβούλιο. Και άμα το συμφώνησαν Γαλλία και Γερμανία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι συμβαίνει αυτό. Πάλι θα βρεθούμε ενώπιον των ανθρώπων και δεν θα έχουμε καμία απάντηση για τους ανθρώπους. Πού είναι η παράγραφος όπου προτείνεται πώς θα βγούμε από κοινού από την κρίση με ανάπτυξη. Αυτό είναι το κενό το οποίο διαψώνουμε εμείς ως ομάδα. Ναι, συμφωνούμε με τους συναδέλφους που θέλουν πιο πολύ μεταρρύθμιση και εμείς το ίδιο θέλουμε πιο έντονη, αλλά τι θα περιλαμβάνει αν δεν είστε διατεθειμένοι να δείτε την ουσία του προϋπολογισμού και να τα βάλετε αυτά στον προϋπολογισμό γιατί να συνεχίσουμε να μιλάμε για Ευρώπη 2020. Είναι κάτι το κενό ήδη από σήμερα. Μπορούμε να το ρίξουμε από τώρα στην ανακύκλωση, εάν δεν θέλετε να μιλήσετε μαζί μας σοβαρά. Εάν δηλαδή θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε παροχημένες γραφειοκρατίες ή στην ενέργεια του μέλλοντος. Δεν έγινε αυτή η συζήτηση. Και αυτό για εμάς είναι το αποφασιστικό. Επίσης δεν θα αποδεχτούμε εμείς δείκτες που θα προκύψουν μετά από την ομοθεσία. Δεν θα σύρετε πίσω σας το Κοινοβούλιο. Επίσης, θα πρέπει να δούμε την απασχόληση και αν αποτελεί σημαντικό κομμάτι του προπολογισμού ή όχι. Σα ευχαριστώ. Τρεμός, ε, Ραμόν, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί, η οικονομική κρίση δίνει την ευκαιρία, μας δίνει την ευκαιρία να προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα εστιαστώ στην δημιουργία μια ενός κοινού νομισματικού, Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Θα, αυτό θα βελτιώνει πολύ το θεσμικό πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Ξέρω ότι το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο για ορισμένε χώρε, αλλά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα συντόνιζε τις πολιτικές κινήτρων των κρατών μελών και θα, είχε, θα έδινε την ευκαιρία στην Ευρώπη να εκδώσει ευρωομόλογα προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τους δικούς της ε, πόρους ε, δεδομένου ότι οι προπολισμοί των κρατών μελών μειώνονται. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα μπορούσε μάλιστα να, μειώσει τις, ε, να βοηθήσει να μειωθούν οι συνεισφορές των εθνικών προπολογισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς ε, αυτονομία στα έσοδα δεν μπορεί να υπάρχει αυτονομία στις δαπάνες. το Ευρωπαϊκό Κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, αντιμετωπίζει όμως το εξής πρόβλημα. Ε, λείπει η πολιτική βούληση και για την ακρίβεια η πολιτική βούληση της Γερμανίας. Στη δεκαετία του 1990 η Γερμανία προώθησε την ε, υιοθέτηση του ευρώ παρόλο τις δυσκολίες που είχε με την επανένωσή της. Κατά την μου η Γερμανία και τώρα θα πρέπει να ηγηθεί ε, μια, μιας προσπάθειας για τη δημιουργία ενός ενού Ευρωπαϊκού Ταμείου. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ήβο Στρέζιτσέτσκ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας την αγροσκελή αυτή συζήτηση, θεωρώ πως ε, αυτοί οι οποίοι έχουν δίκιο είναι αυτοί που λένε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Αφενός υπάρχουν αυτοί που θέλουν μια ισχυρή κοινοτική προσέγγιση και από την άλλη Βεβαίω είναι μειονότητα, είναι αυτοί που θεωρούν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται με διακυβερνητικό τρόπο. Εξού και οι ιδέες περί ευρωπαϊκών φόρων με τον εφημισμό αυτό που χρησιμοποιείται περί καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης. Γι' αυτό μιλάμε για εμπάθυνση της Ένωσης, δηλαδή περισσότερες εξουσίες στην Κομισιόν εις βάρος των κρατών μελών. Είναι Κρίμα που δεν ακούσαμε κάποιον να λέει σήμερα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μειωθούν να μειωθεί ο αριθμός των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να μεταρρυθμιστεί η κοινή γεωρική πολιτική. Ευχαριστώ, Γιούργεν Κλούτε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ η οικονομική διακυβέρνηση όπως αναπτύσσεται εδώ πέρα εστιάζει μόνο στην εξοικονόμηση και στον ανταγωνισμό. Το πρόβλημα το ανέφερε μόλις ο Ισπανός συνάδελφος. Είναι το πρόβλημα του ότι η Γερμανία προσανατολίζεται στις εξαγωγές. Είναι προφανώς το κεντρικό πρόβλημα στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γερμανική πολιτική του ανταγωνισμού λειτουργεί εις βάρος της εσωτερικής ζήτησης στη Γερμανία δεν το συζητάμε αυτό, αλλά και εις βάρος των μισθών. Είναι ανταγωνισμός μισθών. Και ο ανταγωνισμός αυτός των μισθών παράγει στις γειτονικές χώρες, στα συνδικάτα, στους εργαζόμενους τεράστια πίεση. Ούτε η Κομισιόν ούτε η Εκθεσφαίη το αναφέρουν αυτό το θέμα. Μια οικονομική διακυβέρνηση αντάξια του ονόματός της θα έπρεπε εδώ πέρα να επέμβει. Δεν επιτρέπεται να σιωπά. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Γκοζές για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα, κύριε Επίτροπε, το 1968 οι φίλοι του συναδέλφου Πεντήτ έγραφαν στους τοίχους του Παρισιού λόγια, όχι πράξεις. Σήμερα το αίτημα των πολιτών είναι το αντίθετο. Πράξεις και όχι λόγια. Ακούμε πολλά λόγια, αλλά οι συμπολίτε μα δεν βλέπουν ε, αποτελέσματα. Η προθεσμία δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανέρχεται στο ύψο των περιστάσεων. Μαζί πρέπει να, να σημειώσουμε πρόοδο μέσα στο κοινοτικό πράγμα. Και ω προ αυτό θα ήθελα να αναφέρω το ρόλο του Κοινοβουλίου. Και εδώ θα πρέπει να γίνουν προσπάθειε ώστε να σεβαστούμε την αρχή τη συναπόφαση. Ε, επανειλημμένος ο πρόεδρος της Κομισιόν ευχαρίστησε το Κοινοβούλιο αλλά το Κοινοβούλιο δεν είναι εδώ για να παίζει το δεύτερο ρόλο της απλής υποστήριξης ή για να επικυρώνει χωρίς να έχει τη δυνατότητα να συζητήσει τις αποφάσεις που λαμβάνει το Συμβούλιο. Είναι σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο και γι' αυτό πρέπει τώρα να το συνειδητοποιήσουμε και ως προ αυτό η συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση θα είναι μια δοκιμή. Ε, τώρα, Όσον αφορά την επερχομενη διασκεψη συνδιάσκεψη G20, θα πρέπει να παίξει το ρόλο της Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το διεθνές όργανο να μπορέσει και αυτό με τη σειρά του να ενεργήσει και να μην αφήνεται μόνο στα λόγια. Ευχαριστώ. Uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε πολλούς ομιλητές, αλλά ο χρόνος ε, τρέχει και όπως ξέρετε στις 12 έχουμε την ομιλία του Προέδρου. Θα είμαι πολύ αυστηρός με το χρόνο, ζητώ συγγνώμη και τον προτέρων γι' αυτό. Θα χτυπώ το σφυρί και μπορεί να έχετε 5-10 δευτερόλεπτα μετά από αυτό μόλις τελειώνει ο χρόνος σας. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τον ε, συνάδελφο Φέιο που έκανε μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια συμβιβασμού των διαφόρων απόψεων. Συμβιβασμός που χαρακτηρίζει την έκθεσή του. Όμως το συμπέρασμα στο οποίο φτάσαμε είναι ότι το ε, Κοινοβούλιο σε συγκεκριμένα θέματα, όπως και στο θέμα της χρηματοοικονομικής εποπτείας, έτσι και εδώ ε, έχει την δυνατότητα να δράει ενωμένο υπέρ των συμφερόντων των πολιτών μας. Και αυτό θα πρέπει να το, γνωρίσει, να το αναγνωρίσει και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ιδιαίτερα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό δεδομένου ότι αφορά ένα πακέτο έξι προτάσεων για πολλές από τις οποίες το Κοινοβούλιο έχει, διαδικασ... έχει δικαιώματα ε, συνομοθέτη. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μαζί μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου. Ο εισηγητή ε, υπογραμμίζει ορισμένα θέματα που είναι πολύ σημαντικά. Η οικονομική διακυβέρνηση, για παράδειγμα, ε, είναι κάτι παραπάνω από ένα πακέτο κυρώσεων. Η ανάπτυξη και η απασχόληση χρειάζονται ιδιαίτερε πρωτοβουλίε. Πρωτοβουλίε που θα αντιμετωπίζουν τις ε, διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζονται λύσεις για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και τα κρατικά χρέη. Όλα θα εξαρτηθούν από τη δυνατότητα του Συμβουλίου και της ε, Κομισιόν να αντιμετωπίσουν τις προσδοκίες, να απαντήσουν στις προσδοκίες των πολιτών τους. Για ένα λεπτό. Thank you. Σας ευχαριστώ. Καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση χρειάζεται με πρώιμη προειδοποίηση και πρώιμη δράση οι στόχοι για τα κρατικά χρέο έχουν παραβιαστεί χρειάζονται μέτρα και για την Ισπανία και για την Ιρλανδία. Η οικονομία δεν είναι μια ακριβής επιστήμη και δεν αφορά μόνο τους αριθμούς. Η ιστορία μας θυμίζει ότι θα πρέπει ότι μάλλον μια ισχυρή χώρα δεν σημαίνει και ισχυρή οικονομία. Κεντρικοί ε, σκυρώσει και κεντρικό ταμείο δεν είναι επίση οι τοπικέ λύσει, οι τέλειε λύσει. Θα πρέπει να ληφθούν διάφορε αποφάσει ώστε να σωθεί ένα, ένα, ένα κράτο το οποίο μπορεί να αποτελεί μια κέννη απειλή. Όμω ε, η ευρωπαϊκή κεντροποίηση μπορεί να επιφέρει περισσότερου κινδύνου. Εγώ καταλαβαίνω ότι ανησυχούν διάφοροι για τι γερμανικέ συμφωνίε συμφωνίες. Όμως ίσως έχει νόημα κάτι τέτοιο. Αν η αγορά είναι αυτή που δανείζει τα χρήματα, τότε ίσως αυτή θα πρέπει να φέρει και τη ζημιά και όχι ο φορολογούμενος. Ε, Συνάδελφοι, ως συνήθως έχουμε και τα καλά και τα άσχημα στην πραγματικότητα και στο τι κάνουμε. Βεβαίω πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το παρελθόν και τι αιτίε τη κρίση και νομίζω πω η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει κάνει αυτό. Αλλά σήμερα πρέπει να δώσουμε βάση στο μέλλον και στο παγκόσμιο και στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση που είναι για το αύριο. Δεν αφορά μόνο αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Η Ευρώπη δεν υφίσταται σε ένα κενό. Όταν κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε την Ευρώπη το κάνουμε σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο που είναι τελείως διαφορετικό από το 2008 η G20 ήταν ενωμένη για τις διασώσεις πριν από δύο χρόνια αλλά η ομοφωνία αυτή βεβαίως βασίζονταν στο φόβο Σήμερα λοιπόν είναι διχασμένη. Δεν υπάρχει παγκόσμιο κοινό καλό. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που δρούν για την ανάκαμψη και την ε, επανισορρόψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν διορθωτικές αλλαγές που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ο ρόλος των νομισμάτων ως ε, παγκόσμιο μηχανισμό εξορρόψης έχει αυξηθεί πάρα πολύ και βλέπουμε ένα νέο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα με περισσότερους παίκτες. Για να μην έχουμε λοιπόν ασύμετρες προσαρμογές είναι πήγον ένας διάλογος. Το θέμα το οποίο τίθε λοιπόν εάν ε, η Ευρώπη θα έχει τη δυνατότητα να παίξει τον ρόλο της. Οπότε αυτό το οποίο λείπει είναι μία μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης. Με το να μην το κάνουμε αυτό, χάνουμε επιρροή. Υπό τις παρούσες συνθήκες η Ευρώπη δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρώπη δεν πάει καλά, ούτε και ο κόσμος. Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπο Συμβουλή υπογράμμισε πω η παγκοσμιοποίηση απαιτεί δράση σε ευρωπαϊκό και σε διεθνέ επίπεδο αλλά παρατηρώντας τα όσα συμβαίνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο αναγκαζόμαστε να διαπιστώσουμε πως προ... ακριβώς οι συγκεκριμένες δράσεις είναι που λείπουν. Η διάσκεψη της διάσκεψης, οι διάφοροι σπουδαίοι και λιγότεροι σπουδαίοι που θέλουν να, να διευθύνουν επαναλαμβάνουν και παπαγαλίζουν τα ίδια. ενώ βασικό συμπέρασμα της κάθε διάσκεψης κορυφής είναι να ξανασυνεδριάσουμε. Η διεθνής διακυβέρνηση, G20, Καμιά νομική βάση δεν υπάρχει σε, ούτε σε διεθνές επίπεδο και λειτουργεί το σύστημα αυτό εκτός του ΟΗΕ. Οι G20 αυτοδιακήρυξαν την λειτουργία τους. Είναι ένα κλαμπ των ε, πλουσίων, ε, αναδυόμενες χώρες ε, σε δημοκρατίες οι οποίες είναι τόσο πολύ υποδειγματικές όπως η Σαουδική Αραβία. Ο Μάρτιν Σούλτ είπε για το G20 ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο με τις, τα ανακοινοθέντα που δημοσιεύονται μετά από τις ευρωπαϊκές διασκέψεις Κορυφή. Ένα σωρό μάταια λόγια και υποσχέσεις. Ποτέ δεν ακολουθούνται από δράση. Η Ευρώπη ακολουθεί τη γαλλογερμανική διάσκεψη όπου το μυστήριο αυτό ζευγάρι, Σαρκοζή, Μέρκελ, προσπαθούν να μας δείξουν το δρόμο. Ο, Φερχόφστατ μίλησε για καζίνο. Ε, εγώ πάω να πω, βάλτε, μιζάρετε, ε, γιατί τίποτα δεν πάει καλά. Θα πρέπει η Κομισιόν να αυξήσει την ευρωπαϊκή μίζα. Μπα και βγούμε από την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ την συγκεκριμένη κυρία Μπερές και όσους συνεισέφεραν για αυτή την Γι' αυτό το κείμενο το οποίο συζητούμε. Αποτελεί μια συνεισφορά που υπογραμμίζει τις, ε, το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ατμομηχανή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 20 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν μπορούσε κάθε μία από αυτές να δημιουργήσει μία θέση εργασίας η ανεργία θα μειωρόταν πάρα πολύ. Επίση, υπάρχουν και άλλες συστάσεις για οικονομικές στρατηγικές για την ε, αντιμετώπιση κρίση. Η πρώτη ανάγκη είναι η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας αγοράς, ε, χωρίς περιορισμού στον ανταγωνισμό και διευκολύνοντας την ε, πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις επιστώσεις. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ακόμα και επιχορηγήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η δημιουργία, η υιοθέτηση μιας Small Business Act που θα εν, τονίζει τον, με, ισχυρή κοινωνική διάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η καινοτομία επίσης είναι μηχανή της οικονομικής ανάπτυξης και πρέπει να προστατευτεί και να συνδεθεί οργανικά η καινοτομία με τη βιομηχανία. Χρειάζονται καινούριε συμμαχίε ανάμεσα στην βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό τομέα και επίση ε, ένα, εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολισμένο στην αγορά εργασία. Ταυτόχρονα χρειάζονται καινούργια προσόντα για καινούριε θέσει εργασία. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε Κύριε Επίτροπε, ο κύριος Μπαρόζο είπε στην αρχή πως ε, η οικονομική διακυβέρνηση αναπτύχθηκε τόσο γρήγορα ώστε πριν από δύο χρόνια κανείς δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει τα όσα συνέβησαν. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά η ταχύτητα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Πρέπει να είμαστε σίγουροι πως ε, το τρένο ακολουθεί και σωστή πορεία. Και Αυτό νομίζω γίνεται με την ε, ανάλυση της έκθεσης ε, Μπερές. Εδώ πέρα πρέπει να ακούσουμε τον Νομπελίστα, τον κύριο Κρούγκμαν και διαφόρους άλλους ε, αντιφρονούντες που λένε πως εδώ πέρα θυσιάζονται θέσεις εργασίας σε κάποιους βομούς από τις κυβερνήσεις. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ως δείκτη και το επίπεδο ανάπτυξης, γιατί, ε, ανα, απασχόληση, με συγχωρείτε, γιατί θα επηρεαστεί η πραγματική ε, οικονομία και αυτό θα... Και επίσης με απασχολεί αυτό που είπε ο κ. Σόλε Σμιτ. Στην έκθεση της Task Group ε, γίνεται μια έκκληση για μια κοινωνική προσέγγιση προκειμένου να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ο συμβασμός ε, αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ο ειδικό μα συμβασμό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι αφορά το σύμφωνο σταθερότητα, πώ μπορεί να λειτουργήσει, πώ μπορούμε να εξηγιάνουμε του προπολογισμού και ποιοι είναι οι αντικειμενικοί στόχοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σημαντικέ ε, αποφάσεις οι αποφάσεις δε για την ε, πολιτική συνοχή θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί η πολιτική συνοχή θα συνεισφέρει στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την μελλοντική μας ανάπτυξη. Θα πρέπει να δοθεί ένας καινούριος ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και θα μειώνει τα γραφειοκρατικά βάρη. Είμαι σίγουρη ότι οι συστάσεις μας θα οδηγήσουν σε ανάληψη δράση από πλευρά των, της Κομισιόν. δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο. Οι πολίτες μας περιμένουν γρήγορες απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι κάποιοι άνθρωποι μου κουνάνε πολύ χαρούμενα το χέρι. Όμως όταν να τους ε, αντιχαιρετώ σημαίνει πως έχουμε γράψει τα ονόματά τους στον κατάλογο. Δεν χρειάζεται να ζητάτε και από τους υπόλοιπους συναδέλφους να κουνούν τα χέρια τους, να με χαιρετάνε. Δεν σας εγγυώμαι βέβαια ότι όλοι θα μιλήσετε γιατί το, η διαδικασία ΚΑΣΔΙΑ εξαρτάται από το χρόνο που έχουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει διαφορετικά τα κράτη-μέλη. Η διαφορά όμως δεν περιορίζεται εντό των ορίων της Ευρωζώνης όπως θα έλεγαν κάποιοι οικονομολόγοι στο παρελθόν. Ούτε υπάρχει τέλεια συνοχή. Οι χώρες της Ευρωζώνης είναι πολύ διαφορετικές τώρα από όταν εισήχθη το ευρώ και είναι προφανές πως το σύμφωνο σταθερότητας δεν περιέχει τους σωστούς δείκτες. Γι' αυτό η αυτόματη επιβολή κυρώσεων δεν θα έχει αποτελέσματα από μόνη της και νομίζω πως ε, ο αντίκτυπο δεν θα είναι καλό σε όλα τα κράτη-μέλη. Τα οικονομικά κλισέ θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα. Η λύση είναι προφανής. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εναρμονίσουν τις οικονομίες τη, έτσι ώστε να ε, έχουμε τα ίδια αποτελέσματα με τα ίδια μέσα, δηλαδή περισσότεροι Ευρώπη και υψηλότερος προπολογισμό και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ίδιους πόρους. Κύριε Πρόεδρε, η κρίση δεν βρίσκεται στο τέλος της και το βλέπουμε αυτό. Στην Ευρώπη φαίνεται αυτό να αποτελεί πλέον μια κρίση ολοκλήρωσης και αυτό μετά από την ε, ε, συμφωνία της Ντοβίλ που τορπιλίζει την κοινοτική μέθοδο και με δείχνει τελικά ποιοι ε, εξακολουθούν να είναι ισχυροί. Το 2050 νομίζω πως η Ευρώπη θα αντιπροσωπεύει ακόμα το 6-7% του παγκόσμιου πληθυσμού με μια οικονομική δύναμη η οποία θα καταραίει. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να κάνουμε ανταγωνισμό στον εαυτό μας, έτσι θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του διεθνούς ανταγωνισμού ή μήπως θα πρέπει να υπακούσουμε στην κοινοτική πειθαρχία και λιτότητα και να ενεργήσουμε από κοινού για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει Για να το κάνει αυτό χρειάζεται καινοτόμα μέσα η Ευρώπη και η συζήτηση περί των νέων δημοσιονομικών προοπτικών είναι μια καλή ευκαιρία για να τα αναζητήσουμε αυτά. Για τα θέματα ανάπτυξη και έρευνα. εξωτερική υπηρεσία επίση. Τι χρησιμεύει ακόμα μια νιωστή διπλωματική, ένα νιωστό διπλωματικό σώμα τη Ευρώπη που ενώ υπάρχει ήδη κάτι τέτοιο θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο περιθώριο στα κράτη για να το παγιώσουν και να δώσουμε στην Ευρώπη τα μέσα που, έχει, που χρειάζεται ώστε να έχει μια πολιτική που να γίνεται αντιληπτή από τους πολίτες. Μα, το απαιτούν αυτό. Ja, Präsident, äh, ich denke, wenn man der Debatte heute Morgen zugehört hat, merkt man, dass wir in den... Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση μας ε, οδήγησε να διαπιστώσουμε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ε, έχουμε δουλέψει καλά και αυτό δεν χρειάζεται να το κρύψουμε. Ε, μιλάμε για την Επιτροπή για την κρίση, έχουμε δουλέψει πολύ σε αυτήν. Έχουμε 1.600 τροπολογίες στην αρχική έκθεση και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι απόλυτο σωστό διότι η κρίση δεν έχει καθόλου τελειώσει αντιθέτως ε, βλέπουμε ότι η Ιρλανδία μόλις ε, ε, απόφυγε την πτώχευση η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι καλή ως εκ τούτου πρέπει να συνεχίσουν οι οικονομικές αλλαγές και θα πρέπει ήδη να τελειώσει αυτή η διαδικασία θα ήταν ε, ε, λάθος να θεωρήσουμε ότι έχει τελειώσει η διαδικασία και μπορούμε ε, να αποποιηθούμε την εντολή μας. Γι' αυτό και νομίζω ότι είναι αποδεκτή η έκθεση και αυτό άλλωστε φάνηκε στην Ειδική Επιτροπή. Θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε πει ορισμένα πράγματα καλύτερα, αλλά εδώ πρόκειται για μια μεταβατική έκθεση. Οπότε, στο δεύτερο ήμιση Τη της ε, ε, θητείας της Επιτροπής θα συνεχίσουμε την εργασία που έχουμε ξεκινήσει θα δούμε πόσο μπορούμε να τύχουμε στήριξη και στις άλλες επιτροπές για την εργασία την οποία ήδη έχουμε κάνει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα σήμερα το πρωί πολύ προσεκτικά τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε κάπως τα πράγματα, να δούμε ποια είναι τα μέσα που είναι καλά καθορισμένα και καλά ευθυγραμμισμένα στη στρατηγική και την εσωτερική μας ενότητα σαν ευρωπαϊκή κοινότητα. Όσον αφορά τα μέσα, τα εργαλεία, πιστεύω ότι έγιναν βήματα προόδου πάρα πολύ σημαντικά. Πιστεύω συνεπώς ότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι η στρατηγική. Στη στρατηγική αν είμαστε στην ίδια γραμμή. Διότι πάντα μιλούσαμε για σταθερότητα, όμως είναι η ώρα και καθυστερήσαμε μάλιστα να μιλήσουμε για ανάπτυξη. Λοιπόν, όταν μιλάμε για σταθερότητα και θυσία, εγώ συμφωνώ απόλυτα, αλλά ταυτόχρονα εάν δεν βασιστούμε και στην ανάπτυξη μέσω της απασχολήσεως, που είναι κρίσιμο ζήτημα την περίοδο αυτή. Αν δεν το κάνουμε αυτό λοιπόν, ε, δεν θα κάνουμε καλή δουλειά. Πάνω σε αυτό, πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επενθυμίσουμε στον Παρόσο που ήρθε να παρουσιάσει την κατάσταση της ενώσεως εδώ πρόσφατα. Ε, ε, ε λοιπόν, και αναφέρθηκε στη χρηματοστητική αγορά τότε. Σήμερα δεν τον άκουσα να μιλήσει. Θα ήταν σφάλμα ασυγχώρητο αν θέλαμε να καλύψουμε την αναρχία που επικρατεί μεταξύ των κρατών πίσω από την έννοια της επικουρικότητας. Πολύ λίγο χρησιμοποιείται και περισσότερες φορές με κακό στόχο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρινς για 1,5 λεπτό. Eh, Κύριε Πρόεδρε, κύριοι ευρωβουλευτές, ε, ε, ε, εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ε, βλέπουμε ε, τώρα τα αποτελέσματα της κρίσεως και ε, ακόμη και στην Λετωνία, στη χώρα μου, οι πολίτες υποφέρουν. Έχουμε μία μείωση κατά 20% της οικονομίας, η ανεργία έχει εξελιχθεί πολύ ταχαίως και σε μία τέτοια έκτακτη κατάσταση χρειάζονται έκτακτα και ειδικά μέτρα. Τι μέτρα λοιπόν έχουμε λάβει για να επιλύσουμε και να τακτοποιήσουμε τα οικονομικά μας θέματα. Οι πολίτες της χώρας μου έχουν δεχτεί ε, κατά 30% μειώσεις μισθών, έχει αυξηθεί η φορολογία και η οικονομική μας σταθερότητα μπόρεσε να εδρεωθεί. Αλλά ανησυχώ γιατί σήμερα διαβάζω ότι η Γαλλία και η Γερμανία δεν επιθυμούν να ενισχύσουν την ε, ε, οικονομική διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να την αποδυναμώσουν. Αυτό σημαίνει ότι στη χώρα μου οι πολίτες ε, δέχτηκαν τις θυσίες αυτές ανεφλόγου. Υπάρχει μια κατάσταση όπου οι χώρες δεν μπορούν να συνεχίσουν όπως ήταν στο παρελθόν. Θα χρειαζόμαστε η Επιτροπή να έχει πιο σαφή καθοδήγηση. Κύριε ε, Πρόεδρε, θα πρέπει να, ο κύριος Χάκμαρ να δεχθούμε ότι ουσιαστικά η οικονομική κρίση αναφέρεται στην Ευρώπη και ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Στα άλλα μέλη του κόσμου η ε, αύξηση οικονομική είναι σημαντική. Ως εκ αντιμετωπίζουμε μία μεγάλη πρόκληση, δηλαδή να έχουμε ανάπτυξη και να σταθεροποιήσουμε τα δημόσια οικονομικά μας. Οπότε αυτό είναι η ανησυχία μου, διότι βλέπουμε ότι ορισμένοι αρχηγοί κρατών στην Ευρώπη μιλούν για πιο χαλαρούς ή ευέλικτους κανόνες για το σύμφωνο σταθερότητος και ε, προωθούν μία αλλαγή των συνθήκων. Εγώ δεν νομίζω ότι η Ευρώπη χρειάζεται συζητήσει για συνταγματικές αλλαγές. Ε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, ε, το σύμφωνο σταθερότητος με αυτόματες κυρώσεις ισχυρές, να μειώσουμε τα ελλείμματα των προπολογισμών αποτελεσματικά και να μεταρρυθμίσουμε για να ανοίξουμε τα σύνορά μας ε, για οικονομική ανάπτυξη, για μεγαλύτερο ανταγωνισμό και αυτό πρέπει να προωθήσουμε και στο G20 και για, την για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Κύριε Πρόεδρε, στην έκθεση Μπέρες για την οικονομική κρίση την οποία μεταξύ άλλων συζητούμε σήμερα στην παράγραφο 32 επισημαίνεται ότι ορισμένα κράτη μέλη και εδώ υπονοείται σαφώς και η χώρα μου η ελλάδα δεν έχουν επί του παρόντος τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πραγματικά σχέδια ανάκαμψης και όλες οι δυνατότητες επιλογής περιορίζονται μέχρι το 2012 σε περικοπές των δημοσίων δαπανών αυξήσεις της φορολογίας και μείωση του χρέους η θέση αυτή έχει τεράστια σημασία για την ελλάδα μεταξύ άλλων καθώς στο εσωτερικό της χώρας υπάρχουν δυνάμεις που ισχυρίζονται το τελείως αντίθετο. προσωπικά θα ήθελα να υποστηρίξω τη θέση αυτή της έκθεσης μπέρες, καθώς σε χώρες όπου το έλλειμμα και το χρέος είναι πολύ μεγάλα και ακόμη περισσότερο σε χώρες οι οποίες έχουν χάσει την πρόσβαση στη διεθνή αγορά κεφαλαίων η ανάκαμψη περνά αναγκαστικά από τη μείωση των ελλημάτων δεν υπάρχει άλλος δρόμος. αν δεν μειώσεις τα ελλείμματα δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. αν δεν έχεις πρόσβαση στις διεθνείς αγορές δεν μπορείς να πετύχεις ανάκαμψη. είναι ένα πικρό ποτήρι ιδίω για τους πολίτες αλλά πρέπει να έχουμε το θάρρος να λέμε στους πολίτες την αλήθεια. ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. τώρα περνάμε στη διαδικασία του catch the eye Κύριε με βάση το χρόνο που έχουμε αναμένω να μπορέσω να δώσω το λόγο σε περίπου 10 συναδέλφους. Αυτό θα πει ότι περίπου 6 ή 7 δεν θα πάρουν το λόγο, εκτός αν είναι πολύ σύντομοι οι υπόλοιποι. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι είναι η κατάσταση και δίνω τον, τον λόγο όπως τον έχω στο χαρτί μπροστά μου, με αυτή τη σειρά. Ο κύριος Κέλλη, για ένα λεπτό ακριβώς. I will be very strict in this. One minute. Mr. Kelly, one minute. One minute it shall be. Ε, Για ένα λεπτό. Δύο δηλώσει έγιναν το πρωί και εκεί θα στοχεύσω. Η κυρία Ντανίτα Χούπνερ που είπε ότι δεν υπάρχει σε κενό η Ευρώπη και ο κύριο Σαστέλ είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει όλε τι παραχωρήσει μόνη τη. Ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει σκληρή, κυρίω με τι χώρε των G20 και των ΟΗΕ. Είμαστε σε μια θέση όπου έχουμε 11% ανεργία, 20% ανεργία στου νέου, τεράστια δημόσια χρέη και πολλού σε φτώχεια. Και αν οι άλλε χώρε στον κόσμο δεν μοιραστούν το βάρος, εμείς θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα το κάνουμε πλέον. Να επιτρέψουμε στις χώρες μας να μην γίνονται ανταγωνιστικές και να αυξηθεί η φτώχεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, θέλω να πω ότι εντός της Ευρώπης δεν χρειάζεται μόνο να μιλάμε μια φωνή, αλλά να δράσουμε και σαν ένα κορμί. Και το Διοικητικό Συμβούλιο που αυτοδιορίστηκε και επαναφέρθηκε σήμερα το πρωί δεν μπορεί να συνεχίσει ε, να κινείται με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Ε, για ένα λεπτό. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το ότι συντάσσεται μια έκθεση η οποία αφορά ε, την καλύτερη διακυβέρνηση και το πλαίσιο σταθερότητας. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Φέγιο. Είμαι βέβαιος ότι οι νέες πρωτοβουλίες όπως ε, οι δέσμοι μέτρων χρηματοοικονομικής εποπτείας ή το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα αποτρέψουν μελλοντικέ κρίσεις ή τέλος πάντων ε, θα μετριάσουν τα αρνητικά τους αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η βελτίωση του συντονισμού, να υπάρχει καλύτερη προβολή των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης ε, τη σημασία ενός καλού πλαισίου για την οικονομική συνεργασία ε, σε επίπεδο Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών ταπανών που ε, συνδέονται με τις κοινοτικέ αντίστοιχε Σε Αυτή η συνεργασία θα οδηγήσει και στη διενέργεια κοινοτικών οικονομικών αναλύσεων. Περνιώ ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, με λίγα λόγια, καταρχήν μία παρατήρηση για τις ε, προ... Ε, γαλλογερμανικές προτάσεις. Νομίζω ότι πρέπει ε, να αντιδράσουμε θετικά και το λέμε συχνά από το 2007. Δεν υπάρχει πλέον η ατμομηχανή συνδυασμένη της Γερμανίας με τη Γαλλία, αλλά τελικά η πρόταση αυτή έχει και μία χρειά σκλαβιάς, διότι οι προτάσεις αυτές γίνονται για να αποφύγει η Γαλλία βάσει της κακής οικονομικής της υγείας να βρεθεί σε δυσχερή κατάσταση. Πρέπει επίσης να διαπιστώσουμε ότι στις προτάσεις αυτές δεν υπάρχει καμία θετική πρόταση όπως ε, το προωθεί η έκθεση Μπερές για να μπορέσει όντως να υπάρξει μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η κρίση είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο και θα ήθελα συντομία να αναφέρω κάποια σημεία. Στις εθνικές οικονομίες τονίζεται ιδιαίτερα το κριτήριο του δημοσίου χρέους. Και άλλα κριτήρια όμως είναι εξίσου σημαντικά. Το δημόσιο χρέος βεβαίως πρέπει να παρακολουθείτε διότι θα πρέπει τα ελλείμματα να καλυφθούν από οικονομικές δραστηριότητε στο δημόσιο τομέα. Και έτσι όμως ε, και έτσι να προωθηθεί η ανάπτυξη και να μειωθεί η ανεργία. Εμείς εστιαζόμαστε σε στοιχεία που δεν έχουν δημιουργήσει την κρίση. Η ανεργία επιδεινώνει την κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Χωρί σωστέ κοινωνικέ και οικονομικέ πολιτικέ και βελτίωση του οικονομικού τομέα, θα είναι δύσκολο να βγούμε από την κρίση. Και τέλο, κύριε Επίτροπε, επί χρόνια ζητούσα να ασχοληθούμε με το θέμα των φορολογικών παραδείσων. Προτείνω στο μέλλον να έχουμε έναν εκπρόσωπο ε, για τα οικονομικά θέματα. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε έναν ύπατο εκπρόσωπο για τα οικονομικά ζητήματα, όπως έχουμε ύπατο εκπρόσωπο για τις εξωτερικές υποθέσεις. Και ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω. Είναι τροπή που δεν μπορούμε να εκφραστούμε με μία φωνή στις συνεδριάσεις ε, του G20. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά τη Γαλλία, το Σαρκοζή και τον πρόεδρο του G20 στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μία θέση, δηλαδή έναν εκπρόσωπό τη σε αυτέ τι συνεδριάσει, ώστε να μιλάμε μία φωνή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίγκολτ, για ένα λεπτό. Κύριε Ρεν, εχθές το βράδυ όντως ε, ε, υπέφερα για λογαριασμό σας διότι είδα στην συνέντευξη τύπου πως χρειάστηκε να παρουσιάσετε αυτή τη συμφωνία που δεν βασιζόταν μόνο στις δικές σας προτάσεις. Άρα μετά από ό,τι αποκομίσαμε από το εποπτικό πακέτο είδαμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να συνεργάζονται για να επιτύχουν καλό αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα ε, όταν κοιτάμε το έλλειμμα και τις διαδικασίες ελλείμματος καθώς και τις προτάσεις σας σχετικά με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες είναι βασικό για να έχουμε μία σωστή συμφωνία οι ελληματικές χώρες να φέρουν το βάρος των ευθυνών τους κατά τρόπον ώστε να ορθοποδήσει το ευρώ και μπορώ να πω ότι η πλειοψηφία αυτή, αυτού του κοινοβουλίου είναι έτοιμο να στηρίξει τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από δεν έχει θέση η γαλλογερμανική συνεννόηση θέση στο Κοινοβούλιο, έχω κάποιες ερωτήσεις να θέσω στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η ιδέα των ε, επιτοκίων και των καταθέσεων. Ποιος είναι ο λόγος να προσθέσουμε έλλειμμα στο έλλειμμα για την καταπολέμηση του έλλειμματος. Ποια λογική ακολουθείτε. Ένα άλλο ερώτημα που αφορά τη δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας των διεθντικών ταμείων. Ε, αυτό θα έχει σαν συνέπεια καθυστέρηση μέσω μακροπρόθεσμα της ανάπτυξης, αύξηση των επιτοκίων και άρα αύξηση το βραχυπρόθεσμα του ελλείμματος. Πιστεύω ότι θα έπρεπε ίσως να επιβληθούν κυρώσεις κατά της ανοησίας. Thank you, Mr. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Μας υποσχέθηκαν οικονομική ανάπτυξη, αλλά λόγω του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν από τις αναπτυσσόμενες χώρες οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα καταστροφεί ουσιαστικά η βάση της μεταποίησης θέσης εργασίας ο μόνο τρόπο να ανταγωνιστούμε αυτέ τι χώρε είναι να κατεβάσουμε το επίπεδο διαβίωση ε, των εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε την παγκοσμιοποίηση, να προστατεύσουμε του εργαζομένου μα ε, και να είμαστε κατά αυτού του ανταγωνισμού. Βλέπουμε πως οι οικονομίες ε, των κρατών μελών είναι πολύ διαφορετικές. Δεν μπορεί λοιπόν να ε, αρκεί η ίδια συνταγή και για τις 27 χώρες. Θα πρέπει λοιπόν η κάθε χώρα να καθορίσει μόνη της την οικονομική της διακυβέρνηση. Η οικονομική κρίση άλλωστε ξεκίνησε με τις τράπεζες. Αλλά ε, αυτό που έγινε τελικά πρώτα απ' όλα ήταν ότι τρέξαμε να σώσουμε αυτές τις τράπεζες. Πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που κάνουν οι τράπεζε που έχουν στόχο μόνο να προωθήσουν τους δικούς τους τόκους να, κάνουν, να αποκομίσουν κέρδος και όχι να βοηθήσουν τους δικαιούχους, τους πελάτες τους. Mr. Kozlovsky, are you here? Κύριος Κοσλόφσκι. Oh, yes. Mr. Kozlovsky, one minute. Take the floor, lose the floor. Κύριε Κοσλόφσκι, για ένα λεπτό ή θα αρχίσετε να μιλάτε ή θα χάσετε τη σειρά σας. Μίλησα, μίλησα. Έχω μιλήσει κύριε Πρόεδρε, αυτό σας είπα. Έχω μιλήσει στο πλαίσιο του Catch Έχω ήδη λάβει το λόγο, έχω μιλήσει ήδη. Uh, Εγώ είχα τον κύριο Μέσαρο στον κατάλογο. Δεν είστε εσεί ο κύριο Μέσαρο. Τέλο πάντων, το λόγο έχει ο κύριο Μέσαρο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τα προβλήματα και η οικονομική και η κοινωνική κρίση, οι σημαντικότεροι που βιώνουν οι ευρωπαϊκέ οικονομίε. Ε, δημιούργησαν και κάποιε δυσκολίε χρηματοοικονομική ρύθμιση, ιδίω ό,τι αφορά τι πολιτικέ των κρατών μελών. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστέρησε να δώσει απαντήσει και ξέρουμε τι επιπτώσει. Μάλιστα, οι απαντήσει που έδωσαν τα κράτη-μέλη δεν ήταν εναρμονισμένε. Στο μέλλον, λοιπόν, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς εγκαίρως για να υπάρχει ασφάλεια και για να μπορεί να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε συνέχεια ε, στις εργασίες της Ειδικής Επιτροπής εφόσον δεν έχει, πλέον, ε, δεν έχει ακόμη λήξει η κρίση, δεν υπάρχει σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, θα πρέπει να υπάρξουν σχετικές πολιτικές στον τομέα των δαπανών και θα πρέπει να δούμε την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς που είναι ένα στοιχείο ανάπτυξης εξού και η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 είναι σημαντική για την ανάπτυξη, για την απασχόληση. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση για τι μικρομεσαίε επιχείρησει, ε, αλλά και η έρευνα και η καινοτομία επωφελούνται. Ε, η κυρία Παπαδοπούλου για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όντω σε ένα σταυροδρόμι. Η διεθνή οικονομική κρίση συρρήκνωσε την ανάπτυξη, επιδίνωσε την ανεργία, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τα μέτρα διάσωση ήταν θετικά παρά τι σοβαρέ αδυναμίε. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πω απαιτείται περισσότερη κοινοτική αλληλεγγύη και συντονισμό μεταξύ των εθνικών σχεδίων ανάκαμψη το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο απαιτεί από την επιτροπή περισσότερη ευρώπη λιγότερη γραφειοκρατία στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασία περισσότερου οικονομικού πόρου για χρηματοδότηση έργων σε νευραλγικού τομεί πιο ισχυρό ρυθμιστικό εποπτικό και συντονιστικό σύστημα των οικονομικών φορολογικών και κοινωνικών πολιτικών τη ευρωπαϊκή ένωση. υποστηρίζω και εγώ την ανάπτυξη ενό κοινού νομισματικού ταμείου για να ελέγχει αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. τέλο περήφανη για τον κύπριο νομπελίστα χριστόφορο μπισαρίδη καλώ το ευρωκοινοβούλιο να τον καλέσει εδώ να αναλύσει τι απόψει του για αντιμετώπιση τη ανεργία και των σύγχρονων προκλήσεων. Ο κύριος Λάμπερτς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, θα ήθελα απλώς να τονίσω στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο τις τρεις ελλείψεις που παρουσιάζει η πολιτική. Ε, έχουμε έλλειμματα σχετικά με ε, το χρέος και με την προπτική για το 2020. Χρειαζόμαστε πειθαρχία και στα δύο αυτά θέματα διότι απλώς με, την, με το ευχαλόγιο δεν θα μπορέσουμε να να επανορθώσουμε την οικονομία. Επίσης χρειαζόμαστε τα αναγκαία έσοδα, δεν μπορεί να υπάρχει συντονισμός δημοσιονομικός χωρίς να υπάρχει συντονισμός φορολογικός, αυτό είναι το δεύτερο και τρίτον υπάρχει ένα έλλειμμα δημοκρατικό και αυτό με εντυπωσιάζει για τις προτάσεις της Tax Force σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχει καν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην προετοιμασία τη επομένη Συνόδου Κορυφή των G20. Όλοι τα είπαν οι τη αγορητέ όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη, στην ανάγκη ενισχύσεω τη οικονομική διακυβερνήσεω στην Ευρώπη, να ενισχυθεί το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη και να συμμετέχει περισσότερο στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα λοιπόν να παραθέσω εντάχει τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι χώρε μα και που τίθενται και στα μέλη του G20 και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο, πιστεύω, τη επόμενη συνεδριάσεω στον G20, την πρόκληση του πολέμου των νομισμάτων και τη πτυτικότητα των τιμών των πρώτων υλών. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο θέματα είναι εκείνα τα οποία πραγματικά αποτελούν απειλέ για την ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο και δημιουργούν ανισορροπίε πάρα πολύ μεγάλε στον πλανήτη μας θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διοργανωθεί, να, να καταλήξει κοινέ θέσει, να διαθέσει τα μέσα ώστε να μιλά μια μοναδική φωνή στην επόμενη σύνοδο κορυφή των G20 στη Σεούλ και σε επόμενε που ακολουθήσουν και πιο γενικά όσον αφορά το διεθνέ προσκήνιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούχαν για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα της κρίσης ε, εμένουν. Και θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό να υπενθυμίσω το σημαντικό ρόλο της ε, πολιτικής για την οικονομική και την κοινωνική συνοχή. Ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να πω ότι Πρόκειται, οι πολιτικέ αυτέ μάλλον είναι εκ των όν ουκάνευρα προϋποθέσεις. Έχουμε το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης, ε, αλλά με αυτέ τι πολιτικέ θα υπάρξει προστιθέμενη αξία, θα υποστηριχθούν οι προσπάθειε ανάπτυξη οι προσπάθειε για μια αηφόρο ανάπτυξη. Ενώ συγχρόνω θα αποδείξει ότι υπάρχει αλληλεγγύη σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να γίνουν σημαντικέ επενδύσει στον τομέα των υποδομών, είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε για τι μεταφορέ, είτε για τι επικοινωνίε. Χρειάζεται να υπάρξουν σημαντικέ επενδύσει και αυτοί οι πόροι πρέπει να βρεθούν από διάφορες πηγές και με τις συμπράξεις εταιρικού, ε, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ άλλων. Βέβαια ε, δεν αξιοποιούνται πλήρως μέχρι τώρα τέτοια εργαλεία. Η κυρία Ντάτη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον Διέγκο Φέγιο, τον εισηγητή για την ε, φιλόδοξη πρότασή του και την εξαιρετική έκθεση, διότι το Κοινοβούλιο έχει τη σωστή θέση σε μια σημαντική συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και άλλωστε η ελληνική κρίση έδειξαν ε, ποιες είναι οι αδυναμίες οι οποίες ε, υποθάλπουν στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός για να επιλύουμε τέτοια προβλήματα και γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε το σύμφωνο σταθερότητος και ε, ε, αναπτύξεως και αν θέλουμε να εξηγιάνουμε την κατάσταση των δημοσιονομικών καταστάσεων των χωρών πρέπει να περιοριστούμε αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η οικονομική κρίση συγκλώνησε τους πάντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φτώχεια γίνεται όλο και πιο αισθητή στα κράτη-μέλη. Είδαμε επίση ότι τα εθνικά οικονομική οικονομικής ανακάμψεως ήταν, πάρα πολλά, ήταν ανίσχυρα, ασυντόνιστα. Κάποια κράτη-μέλη δεν είχαν τη δυνατότητα να ετοιμάσουν κάποια σχέδια οικονομική ανακάμψης που θα επέτρεπαν να εφαρμοστούν μέτρα οικονομικά που θα ήταν αναγκαία διότι οι χώρες υποχρεώθηκαν να κάνουν οικονομίες, να μειώσουν τις δαπάνες, να συμμορφωθούν ε, όσον αφορά τις επιταγές του δημοσίου χρέους. Όλα αυτά ε, κατά των συμφοριών των πολιτών συνέβησαν. Παραδείγματος χάρη, οι γυναίκε απειλούνται περισσότερο και μπορεί να βρεθούν στη φτώχεια τη χειρότερη δυνατή. Οπότε ήρθε η ώρα ε, να μάθουμε κάποια πράγματα από την κρίση, να αρχίσουμε να συντονίζουμε τις δραστηριότητέ μας και να εφαρμόσουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς. Σας ευχαριστώ. Λεπτό, έχετε ε, τα χρηματιστήρια μπόρεσαν μόλις να ρυθμιστούν και βλέπουμε ότι ε, δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας διότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από την Κίνα. Χρειάζεται λοιπόν μία επέμβαση η οποία επιβάλλεται από την παγκοσμιοποίηση διότι ε, οι Κινέζοι θέλουν να στηρίξουν τις εξαγωγές τους, οι που τα δικά τους προβλήματα και όλα αυτά είναι εις βάρος όλων των χωρών και γι' αυτό θα πρέπει να αποτελέσουν βασικό θέμα εις ε, την συνεδρίαση των G20 διότι ε, υποβαθμίζουμε σημαντικά προβλήματα τα οποία στρεβλώνουν τις αγορές ε, που θέτουν σε κίνδυνο όλες τις χρηματαγορές του κόσμου. Γι' αυτό και θα πρέπει να προβλέψει κανείς σε μία φορολόγηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών ε, την συνάντηση κορυφής. Ας την γιατί Ευχαριστώ ε, τον, ε, τους συναδέλφους και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε δύο-τρία θέματα. Καταρχάς ό,τι είπε ο κύριος Ντίλ είναι πολύ σωστό για να αναθεωρήσουμε την πολιτική συνοχή θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της πολιτικής να δούμε ε, τι έχει γίνει από την διεύρυνση και να δούμε τι μπορεί ε, να ε, χρησιμοποιηθεί από τα διάφορα ταμεία και να κάνουμε έναν απολογισμό αντικειμενικό για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε για το μέλλον. Επίσης πολλοί αναφέρθηκαν στην εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της ε, παγκοσμίου διακυβέρνησης που είναι πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίω κάποια στιγμή όπου ξαναξεκινά ένας πόλεμος των τιμών συναλλάγματος Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν συντονισμένες κινήσεις εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι εσωτερικά και προς τα έξω στις εκπροσωπήσεις μας. Διότι όπως ελέγχθη το G20 δεν είναι ίσως μία λύση στην οποία να αποβλέπουμε τελικά όπου ο καθένας θα έχει τη σωστή του θέση και θα μπορέσει να ισχύσουν οι αρχές διαιτησίας τις οποίες χρειαζόμαστε. Ε, στον ΟΗΕ όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας εχθές θα πρέπει να επιζητήσουμε την ε, οδό για την επίλυση των προβλημάτων στο μέλλον. Και τέλος σχετικά με αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος κύριος Λομπέρ όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις. Εμείς ζητάμε στην έκθεσή μας η Επιτροπή να εξετάσει ετήσια τις ανάγκες των δημοσίων και ε, ιδιωτικών και να έχουμε ένα τυφλοσούρτι που να μας επιτρέπει να προσβλέπουμε μακροπρόθεσμα σε μια στρατηγική προς όφελος των πολιτών που θα βασίζεται σε μια διάρκεια των οραμάτων μας και σε μια συνεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ. Σφέιο, για Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους ε, για τις παρεμβάσεις τους, ακόμη και αυτή τη στιγμή που ολοκληρώνεται η συζήτηση. Πλέον έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε από τα λόγια στα έργα από τώρα και μετά και μετά την ψηφοφορία που ελπίζω να έχει θετική έκβαση το Κοινοβούλιο θα έχει πλέον ε, μία δική του θέση σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Θα υπερασπιστούμε λοιπόν ε, το κοινοτικό πνεύμα, την μεγαλύτερη διαφάνεια και προβολή. Θα υπερασπιστούμε τελικά ένα οικονομικό μοντέλο που περιλαμβάνει έναν στόχο, στόχο των 27 κρατών μελών για ανάπτυξη, με καλύτερο συντονισμό μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μεγαλύτερη οικονομική και νομισματική ένωση. Για να, για να υποστηρίξουμε λοιπόν μια πιο αλληλέγγυα, πιο έτοιμη και πιο αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρώπη όπου όλοι έχουν μεν διαφορετική φωνή αλλά ε, εκφέρουν ένα κοινό λόγο όπου λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις ε, και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρώπη της Οικονομικής Διακυβέρνησης δεν είναι η Ευρώπη των ε, διασκέψεων κορυφής σε διμερές επίπεδο παραδείγματος χάρη. Είναι πολυμερής. Επίσης ακούγεται η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών θα ήθελα να τονίσω και το θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να έχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια για το θέμα αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένα δικό μας όραμα για την μακροοικονομική εποπτεία που θα πρέπει να ασκήσουμε απέναντι στα κράτη-μέλη. Να έχουμε τη δική μας φωνή σε ό,τι αφορά τον τρόπο συμπερίληψης ε, της στρατηγικής 2020. Ε, θα πρέπει επίσης να αναλύσουμε με προσοχή ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξη. Το Κοινοβούλιο έχει διατυπώσει προτάσεις ε, που διαφέρουν από τις προτάσεις των άλλων θεσμικών οργάνων. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή όλοι μαζί με δύναμη να υποβάλουμε τι προτάσει αυτές. Στον όνομα τη Επιτροπή, ο κύριο Ρεν για πέντε λεπτά. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συζητητές κυρία Μπέρες Φεγιό και τα αξιότιμα μέλη για την ουσιαστικότητα αυτή συζήτηση που έλαβε χώρα. Καταλαβαίνω ότι το βάρος των παρεμβάσεων αντιστοιχεί στη σημασία των προσυζήτηση θεμάτων. Έχω κάποια σχόλια και απαντήσεις και παρατηρήσεις όσον αφορά τη συζήτηση και τις εκθέσεις. Θα ξεκινήσω με το διεθνές προσκήνιο. Στην παγκόσμια οικονομία οι μεγάλες ανισορροπίες και οι κρίσεις αρχίζουν και αναφαίνονται απειλώντας την βιώσιμη ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Άρα είναι ουσιαστικό, σημαντικό, στη Διπουργική των G20 αυτή την εβδομάδα και Σύνοδο Κορυφή σε 15 μέρες, να γίνει συντονισμό σε διεθνές επίπεδο για να εξισορροπηθεί η παγκόσμια ανάπτυξη. Όλες οι χώρες πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Οι χώρες πλεονάσματο, ενισχύοντας την εσωτερική ζήτηση και οι χώρες οι ελληματικέ, εστιαζόμενε επί των εξαγωγών και τη ανάπτυξη των εξαγωγών. Αφορά εκατομμύρια θέσει απασχόληση στην παγκόσμια οικονομία αυτό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για ισχυρό και σταθερό διεθνές ματοστικό σύστημα όπου οι ισοτιμίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις θεμελιώδεις αρχέ τη οικονομικέ. Είναι ουσιαστικό στοιχείο αυτό. Είναι βασικό στόχος των G20 η εξισορρόπηση της παγκόσμιας ανάπτυξης υπέρ μια μιας παγκόσμιας και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Για τους ίδιους λόγους είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει και να μεταρρυθμίσει τη δική της οικονομική διακυβέρνηση. Οι εκθέσεις που συνετάχθησαν από την κυρία Μπερές και τον κύριο Φεγιό αποτελούν σημαντική συνεισφορά προς αυτό το σκοπό και οι νομοθετικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη στιγμή που θα εγκριθούν θα αποτελέσουν κβαντικό άλμα προ μια εύρυθμη λειτουργία τη ενώσεω και προ μια λειτουργούσα οικονομική ένωση. Ετέθησα να ρωτήσω να απόψει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά του τόξου και του τους φόρους και τους δασμούς επί των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Το συζήτησα αυτό με τον πρόεδρο Μπαρόσο και θεώρησε ότι θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε σχετικά τη θέση μας διότι ε, έγιναν κάποιες συγκεχημένες δηλώσεις σχετικά με το ζήτημα. Είμαστε εν μέσω θεμελιώδους μεταρρυθμίσεως του δικού μας χρηματοπιστωτικού συστήματος και πρέπει να παραμείνει αυτή η ορμή και η όθηση και στο πλαίσιο των G20. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση Πρώτα απ' όλα για ένα τέλος σταθερότητας ή ένα δασμό τραπεζικό, ένα φόρο τραπεζικό, τόσο ώστε ο τραπεζικός και ο χρηματοπιστωτικός τομέας να συμμετέχουν στο, στις δαπάνες και στο κόστος που δημιουργείται από την κρίση και για μελλοντικές επιλύσεις κρίσεων. Αυτό έχει υποβληθεί σαν πρόταση ε, και θα εφαρμοστεί και εφαρμόζεται κάτι μέλη. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θέλει ο χρηματοπιστωτικός τομέας να παίξει ρόλο στην κάλυψη του κόστους της κρίσης και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμευτεί να πιέσει για έναν φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Τρίτον, εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ως επιλογή για ιδίους πόρους στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω μια πρόταση. Σύμφωνα με αυτή, ο χρηματοστοτικός τομέας σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχει οικονομικά μέσω του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Προτείναμε ένα τέλος σταθερότητας, έναν φόρο τραπεζικό και θέσαμε αυτό το φόρο των χρηματοστοτικών συναλλαγών σαν πηγή ιδίων πόρων και έχουμε δεσμευτεί τρίτον να πιέσουμε για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην έκθεση του κ. Φεϊό εμπεριέχεται μια πρόταση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη σύσταση ενός μονίμου μηχανισμού για την πρόληψη κρίσεων και για την ε, επίλυση κρίσεων θα πρέπει να έχει δύο στοιχεία, να εμπεριέχει δύο στοιχεία. Να είναι δυσδιάστατη η προσέγγιση. Πρόληψη της κρίσης πρέπει να υπογραμμιστεί αυτή η πτυχή και λύση των κρίσεων. Καλύτερα κανείς να είναι ασφαλής και να προβλέπει παρά να διορθώνει. Όσον αφορά την επίλυση των κρίσεων, τον Μάιο ήδη είχαμε δηλώσει ότι χρειάζεται ισχυρό πλαίσιο τη διαχείριση των κρίσεων για την Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει σχετικές προτάσεις για έναν μόνιμο μηχανισμό επιλύσεως διευθετήσεως κρίσεων. Θα το κάνει εν ευθέτω χρόνο. Κάποιες γενικές αρχές διεφάνισαν. κυρίως ότι η πρόληψη, η πρόληψη και η επίλυση των κρίσεων θα πρέπει να είναι αλληλένδετα ζητήματα και οδήποτε οικονομική αρρωγή θα πρέπει να ε, χορηγείται υπό συγκεκριμένου αυτηρού όρου. Ένα τέτοιο μόνιμο μηχανισμό πρέπει να ελαχιστοποιεί τα διάφορα ηθικά προβλήματα και να παρέχει κίνητρα για τα κράτη-μέλη για να ακολουθούν μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική και φορολογική πολιτική και να δίνει κίνητρα και στους επενδυτές να ακολουθούν υπεύθυνες πρακτικές δανειοδότησης. Ο κύριος Σμιτ πρότεινε μια τροπολογία. Αφορούσε την εθελούσια συμμετοχή κρατών μελών που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη στο σύστημα κυρώσεων. Στην πρώτη φάση προτείνουμε, όπως ξέρετε, ένα καθεστώς για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Σε δεύτερο στάδιο και για τα 27 κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποστηρίξει την τροπολογία που έχει σαν στόχο Συμμετοχή των κρατών μελών που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη στο καθεστώς κυρώσεων επιθελουσίας βάσεως. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σημειώσαμε ικανοποιητική πρόοδο στα πλαίσια της ομάδας κρούσης και πετύχαμε σύγκληση όσον αφορά τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβερνήσεως. Κυρίως εστιαστήκαμε στην πρόληψη και στις διάφορες δράσεις πρόληψης, τονίζοντας τη βιωσιμότητα του χρέους. Κύριε Επίτροπε, να σας διακόψω, λέει ο Πρόεδρος, και να ασχοληθούμε με μικροοικονομικές ανισορροπίες και να έχουμε αποτελεσματικό μηχανισμό για να επιβάλλουμε τα μέτρα. Προσπαθώ να βοηθήσω, λέει ο Πρόεδρο, κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, να μην το επαναλαμβάνω αυτό κάθε φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Παρακαλώ να πάρετε τι θέσει σα ήσυχα και μη συζητάτε μεταξύ σα. Και κύριε Επίτροπε, μπορείτε να συνοψίσετε, γιατί πρέπει να μιλήσει και το Συμβούλιο, αν έχει την καλοσύνη. Ευχαριστώ, λέω ο κύριο Επίτροπο. Έχω συνηθίσει την κατάσταση. Σα ευχαριστώ που με βοηθήσατε. Και συνεχίζω και οδεύω προ τα συμπεράσματά μου. Και θα ήθελα να τονίσω ότι παρόλο που υπήρξε σύγκληση απόψεων σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπήρχε σύγκληση στην ομάδα κρούση, στην Task Force, τώρα ξεκινά μόλις η κανονική νομοθετική διαδικασία. Μέχρι τώρα είδαμε την αρχή. Ίσως είμαστε στο τέλος της αρχής. Τώρα όμως αρχίζει η πραγματική νομοθετική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν συνομοθετικός φορέας έχει κρίσιμο και αποφασιστικό ρόλο να παίξει. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας και καλούμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι να καταλήξουν σε νομοθετικές αποφάσεις, ούτως ώστε να έχουμε το νέο σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2011 όταν θα γίνει ο νέος μεγάλος γύρος αξιολογήσεως της αποτελεσματικότητας των δράσεων. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ε, είναι πραγματικά θέμα αξιοπιστίας αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα της ενισχύσεως της οικονομικής διακυβερνήσεως και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πράγματι, η κοινοτική μέθοδος είναι αυτή που κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί και να πετυχαίνει αποτελέσματα. Σας άκουσα προσεκτικότατα. Εκτιμώ την αφοσίωσή σας στην κοινοτική μέθοδο. Ξεκινώντας από την παρέμβαση του κυρίου Ντόιλ, του κυρίου Σούλτς, του κυρίου Βερχόφστατ και του κυρίου Κονμπεντίτ, παρόλο που δεν μπορώ να είμαι τόσο καλός ρήτορας. Εν πάση περιπτώσει όλοι μαζί ας αποδείξουμε εκ νέου ότι η κοινοτική μέθοδος μπορεί να δώσει αποτελέσματα και τώρα θα πρέπει να πετύχει τους στόχους της. Το νέο σύστημα της οικονομικής διακυβέρνησης, δηλαδή, και ας συμπληρώσουμε την ισχυρή νομοθετική ένωση με ισχυρή οικονομική ένωση, ούτως ώστε να έχουμε μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση. Σας ευχαριστώ. finally the... Σας ευχαριστώ. Και εν τέλει εκ μέρους του Συμβουλίου κύριος Σαστέλ. Κύριε Πρόεδρε, πολύ γρήγορα. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω καταρχάς εκ μέρους του Συμβουλίου τους δύο εισηγητέ, την κυρία μπερέ και τον κύριο Φέγιο, που συμβολίζουν τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι αυτό. Να πω επίση ότι καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλύσει τάχιστα και με βάση την αρχή της συναπόφασης τι ε, πρωτοβουλίες ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, τι πρωτοβουλίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να έχουμε πραγματικά ε, στην ε, πράξη την εφαρμογή μιας Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης. Νομίζω ότι το Συμβούλιο είναι στη διάθεση του Ευρωκοινοβουλίου για να έχουμε απτή πρόοδο στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Το πολύ η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα σήμερα στις 12.30.